Γκέρενς επί του θέματος αυτού. La Commission euh, souhaite euh, nous faire Θέλει η Επιτροπή να μας πει κάτι. Έχει κάποια ανακοίνωση ή παρατηρήσεις. Ο κύριος Πίτερ Κρέκ Μακκουέιτ ή η κυρία Κάτριν uh, floor. Ευχαριστώ πολύ. Είναι συνάδελφος εδώ για να λάβει το λόγο. Ε, μπορείτε να περιμένετε 10 λεπτά να καθίσει. Monsieur Rodeschauser, je vous donne la parole pour la dernière fois. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου παρέχετε λίγα λεπτά σήμερα το απόγευμα για να πω δύο λόγια σχετικά με μια πενταετή εμπειρία καθοδόν προς την πολιτική της ανάπτυξης. Ελπίζω πως ε, μπορέσαμε να προχωρήσουμε την ε, θεματολόγιο το αναπτυξιακό σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουμε εδώ έναν κατάλογο από ανακοινώσεις και συζητήσεις που είχαμε με το Κοινοβούλιο. Θα μου χρειαζόταν τουλάχιστον μισή ώρα απλά και μόνο να απαριθμίσω τις σχετικές πρωτοβουλίε ε, δεν θα το πράξω, αλλά θα ενθυμίσω ότι στην αρχή εργαστήκαμε σημαντικά επί της κρίσης, υπήρξε τότε η απαρχή της οικονομικής κρίσης και ε, η Κομισιόν μπόρεσε να κινητοποιήσει περαιτέρω κονδύλια για την ε, υπέρβαση αυτής της κρίσης, κρίσης της διατροφικής κλπ. Για της ανθρωπιστικής δύο για να ε, αντιμετωπίσει την κρίση στις ε, χώρες εταίρους και αυτό το πράξαμε σε στενή συνεργασία μαζί με το Κοινοβούλιο. Εργαστήκαμε επίσης ε, για το θέμα της συνοχής των κοινωτικών πολιτικών, την αναπτυξή τους. δουλέψαμε πολύ το θέμα της επιστήμης ασφάλειας και μπορέσαμε μαζί να πετύχουμε σημαντικούς ε, στόχους της χιλιετίας. Εν τω μεταξύ φτιάξαμε ένα ε, track record το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε με υπερηφάνεια. Επίσης <clears throat> είδαμε την ατζέντα ε, Πώς οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που ανέλαβε τις ε, περισσότερες πρωτοβουλίες ε, σχετικά με το θέματα περιορισμού του κατακαιρματισμού της βοήθειας και αυτό το, θα το σε μια εβδομάδα στο Μεξικό σε μια διάσκεψη για την συνέχεια της της, της βοήθειας. Τώρα για την ατζέντα περί των αλλαγών υπήρξαν πολλές συζητήσεις και δώσαμε κάποιες γραμμέ σαφείς και τέλος κατορθώσαμε να εισακουστούμε και να συμφωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το τι θα πρέπει να κρατήσουμε, τι όχι. Ο κ. Πίμπαξ επίσης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπόρεσε να εξευρεθεί ε, μια συμφωνία. Εξετάσαμε επίσης το ζήτημα του προπολογισμού που αφορά στην χρησιμοποίηση του συστήματος ε, αναχώρα. Και επίσης νομίζω ότι ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το μετά 2015 που επηρέασε σημαντικά τις συζητήσεις στη Νέα Υόρκη. Αυτά για να αναφέρω μερικά μόνο ζητήματα επί των οποίων ήμασταν πολύ προχωρημένοι. Εν τω μεταξύ τα πράγματα άλλαξαν, ο κόσμος άλλαξε ήταν, ε, υπάρχουν χώρες που έφτασαν σε ένα ε, ε, επίπεδο διαβίωσης ικανοποιητικότερο. Αυτό μας οδήγησε στην διαφοροποίηση για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταλήξαμε στη συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ήταν ικανοποιητική αυτή η συμφωνία για όλες τις πλευρές. Επίσης, ομού και με τη βοήθειά σας διαπραγματευτήκαμε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο μπορούμε να είμαστε ε, περήφανοι. Είμαστε η μοναδική ε, πολιτική που δεν ε, έτυχε περικοπών. Χάρη στη βοήθειά σας έχουμε έναν προϋπολογισμό ιδιαίτερα ικανοποιητικό και άνετο, ότι δεν φτάνουμε στο 0,7%. Ίσως να είχαμε είμαστε λιγότερο επιτυχείς σε θέματα των μη διακρίσεων και επίσης ε, της απάνθρωπης ε, μεταχείρισης, κάτι το οποίο συμβαίνει δυστυχώς σε μερικές ε, χώρες εταίρους. Εδώ δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Θεωρώ πως παρά τις έντονες συζητήσεις που είχαμε, και τις επικρίσεις που ακούσαμε από κοινού προχωρήσαμε την θεματολόγιο το αναπτυξιακό και με τις πρόσφατες ε, συμφωνίες για την περίοδο των μελλοντική μπορώ να πω από πλευράς Κομισιόν ότι η συμφωνία για το δημοσιονομικό πολιτές πλαίσιο δώσαμε ένα νέο ρόλο του Κοινοβουλίου στην αναπτυξιακή πολιτική ζήτηση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα Ξέρω πως συζητήσατε για τον στρατηγικό διάλογο που αποτελεί κομμάτι αυτής της πολιτικής, αλλά μας έδωσε ε, κάποιες νέες θέσεις του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ήταν πρωτοπόρος σε συζητήσεις, επηρέασε τις ε, διαπραγματεύσεις που κατ' εμάς διεξήχθησαν ικανοποιητικά και από πλευράς Κομισιόν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει. Θα περιοριστώ σε αυτά τα λόγια, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα και τα μέλη τη για τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και μπορέσαμε από κοινού να κάνουμε πράγματα που από μόνοι μας θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόντισάουερ ιδιαίτερα ευχάριστο να κλείνουμε τις εργασίες μας τις πενταετίας κοιτάζοντας προς τα πίσω και βλέποντας ε, ότι η δουλειά μας εστέφθη από επιτυχία. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο σημείο 8 της Μεσσίας Διατάξεως ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των γάμων ανηλίκων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρώτο σημείο που θα μας απασχολήσει είναι πολύ λεπτό ζήτημα και ιδιαίτερα ανησυχητικό διότι πρόκειται για γάμους ανηλίκων στις αναπτυσσόμενες χώρες και στον τρόπο αντιμετώπισης ολοκληρω... με τρόπο ολοκληρωμένο αυτού του φαινομένου. Έχουμε την χαρά να βρίσκεται ανάμεσά μας η μη κυβερνική οργάνωση που είναι αρμόδια για το ζήτημα και θα συζητήσουμε μαζί τους ε, η κυρία Τάνια Κόξ και την καλωσορίζω. Σας δίνω το λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε τη μελέτη πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να σας παρουσιάσω το ζήτημα των γάμων ελίκων από πλευρά του Plan International. Αυτό το θέμα είναι, μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές εδώ και κάποια χρόνια. Ε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, η γάμη ενηλίκων είναι κάτι που αφορά το, όλη την ανθρωπότητα ιδιαίτερα στην Αφρική, η Νίγηρας, Τσάντ, αλλά και στην Νότια Ασία, το Μπαγκλαντέ, στην Ινδία, αλλά ε, συμβαίνουν και παντού, παντού αλλού, συμπεριλαμβάνοντας και της Ευρώπης. Όταν μιλάω για τους γάμου ανελίκους, μιλάω για μια ένωση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, των οποίο ε, τουλάχιστον ένας εκ των δύο είναι κάτω των 18 ετών. Οι γάμοι ανηλίκων αφορούν ιδιαίτερα τις γυναίκες, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τα αγόρια. Θα μιλήσω ιδιαίτερα για γυναίκες, για κορίτσια στην ομιλία μου, διότι δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή στα αγόρια μια τέτοια πολιτική. Έχει όμως τεράστιες συνέπειες στα κορίτσια. Ε, γάμεν ηλίκων που αφορούν γυναίκες οι οποίες, κορίτσια μάλλον, που είναι αδύναμα και είναι, ζουν στο περιθώριο. Ζουν σε φτωχές ε, περιοχές, ε, δεν είναι ε, μορφωμένες, καλλιεργημένες κλπ. Οι 25% των κοριτσιών από φτωχές οικογένειες ε, ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, έναν γάμο όντας ανήλικες. Μία στις τρεις στα κορίτσια στις αναψούμενες χώρες, σε πολλές χώρες παντρεύονται πριν να συμπλούσουν τα 18 χρόνια. Περίπου 90 εκατομμύρια γυναίκες γίνονται νύφες, ε, θα γίνουν νύφες μεταξύ σήμερα και το 2020. 40, 40 εκατομμύρια, εκατομμύρια συγγνώμη, κορίτσια ετησίως. Και επιπλέον 140 εκατομμύρια θα μαντρευτούν ανάμεσα στο 2020 και το 2030. Αυτά τα στοιχεία είναι πάρα, πολύ σοβαρά. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω λίγο για τους γάμους ανηλίκους και τις αιτίες. Γιατί αν δεν βρούμε, δούμε τις αιτίες δεν θα μπορέσουμε να τους αποφύγουμε χωρίζουμε τους εμπλεκόμενους σε δύο. Πρώτον, θέμα ίσων και θύμων και φτώχεια. Τώρα σε ό,τι φορά τα ίση και έθιμα, κοινωνικοί κανόνες οδηγούν την ε, ανισότητα των, ανάμεσα στα, σαφίλα. στα φύλλα. Οι γυναίκες και κορίτσια αξιολογούνται πολύ λιγότερο από ότι οι άνδρες και τα αγόρια σε πολλές κοινωνίες. Για το λόγο λοιπόν αυτό θεωρείται ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτια, δεν μπορούν εύκολα να βρουν εργασία διαφορετικά από αυτήν ε, που να αφορά την καλλιέργεια της γης. Τα κορίτσια είναι ε, η πρώτα, <clears throat> τα πρώτα άτομα τα οποία καταλείπουν τις ε, σπουδές Παραδείγματο χάρη, τα κορίτσια μπορούν να παντρευτούν σε ηλικία κάτω από 18 ετών σε 46 χώρες απλά και μόνο μέσω της έγκρισης των γονιών. Επίσης πολλά κράτη αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια για την επιβολή του νόμου. Στο Μπαγκλαντές έχουν ένα νόμο που απαγορεύει από το 1929 το, το γάμα ανηλίκων αλλά βρίσκεται στην πιο υψηλή θέση σε ό,τι γάμους του Σε ορισμένε περιπτώσεις οι γονείς ε, θέλουν να παντρέψουν τα σκόρες τους για να τις ε, αποτρέψουν από το να πέσουν θύματα σεξουαλικής βίας. Μια δεύτερη αιτία είναι η ένδια, η οποία οδηγεί αλλά είναι και συνέπεια των γάμων ελίκων. Το συνήθως οι κοπέλες αντιμετωπίζονται ως βάρος για την οικογένεια. Και επειδή συνήθως και, και αν παντρευτεί η κοπέλα μπορεί να αποτελέσει ένα κάποιο εισόδημα για την οικογένεια. Και όταν έχουν εγκαταλείψει το σχολείο τα κορίτσια, είναι πολύ πιο εύκολο να παντρευτούν. Όταν παντρευτούν, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να επιστρέψουν στα σχολιά και άρα να βελτιώσουν περαιτέρω την ζωή τους. Και και φυσικά το να γίνει μητέρα έχει επίδραση και στην επόμενη, την υπόλοιπη ζωή της. Και η κοινωνική κανόνη λοιπόν και η φτώχεια παίζουν ρόλο. Ένα, ε, ένα παράδειγμα τώρα για την Αιθιοπία και τον Μπαγκλαντές είναι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κλιματικής φύσης, ε, η μία με την ξηρασία και η άλλη με τις πλημμύρες. Ε, ε, το αντιμετωπίζουν αυτό οι γονείς τους μια στρατηγική επιβίωση δικής τους. Όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παραμείνουν στα σχολεία και περάσουν μετά στην περαιτέρω οι γυναίκες, τότε λιγότερο πιθανότητε έχουν να παντρευτούν μικρές. Ο αριθμός των παιδιών που γεννούν οι γυναίκες ε, και όσο περιορίζεται τόσο πιο καταρτισμένες είναι οι γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να ασφαλίσουμε όλα τα κορίτσια να έχουν πρόσβαση σε ε, εκπαίδευση, σε ασφαλές, ε, κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Ε, ένα πλεονέκτημα που έχουν τα κορίτσια που μένουν ε, πιο πολλά χρόνια στην ε, σχολείο και στην μετέπειτα εκπαίδευση είναι το θέμα της αντιμετώπισης περιπτώσεων ε, αντιμετώπιση μάλλον των, του προβλήματος του, του γάμου ανηλίκων. Τι λοιπόν συμβαίνει αν ε, τα κορίτσια παντρευτούν νέα. Πέραν από την ψυχολογική ή την συναισθηματική ε, ε, αντίδραση υπάρχουν και άλλα δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι, είναι τα θέματα τον της υγείας και τη σεξουαλική βία. Όταν ένα κορίτσι παντρεύεται σε μικρή ηλικία, δεν, το κορμί της δεν είναι έτοιμο για την ε, αναπαραγωγή. Και το επίση δεν είναι σε θέση να ε, διατηρήσει μια ακίηση. Αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο θανάτου. οι κοπέλες ηλικία μεταξύ 15 και 19 έχουν διπλάσιο κίνδυνο να αποβιώσουν κατά τη διάρκεια της από ότι τα κοπέλες ηλικία 20 με 25. Επίσης τα παιδιά που γεννούνται από κορίτσια έχουν υψηλά ποσοστά θρησιμότητας. Το Plan International βγει σε τρία επίπεδα. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει την Ινδία, το Μαγκλαντές και το Νεπάλ. Αυτά είναι τρεις χώρες ε, στην ε, Ασία με το υψηλότερο ποσοστό γάμων ανηλίκων. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουν οι, οι οικογένειες τα επιπτώσεις από έναν γάμο ανήλικου κοριτσιού και αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι συχνά οι οικογένειες παντρεύουν τις ε, κόρες τους ε, προς το ίδιο συμφέρον, να δηλαδή τις προστατεύσουν. Αυτό που είδαμε είναι πως ε, θα πρέπει να δημιουργήσουν κάποιες λέσεις κοριτσιών και παιδιών για να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους καλύτερα και να μπορέσουν να διαφωνήσουν με τις θέσεις των γονιών τους. Και είναι δυνατόν, είναι δυνατόν οι γονείς να αλλάξουν άποψη χάρη στις προσπάθειες που καταβάλουν τα παιδιά τους. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις πρώτα για να προωθήσουμε νομοθεσία και την επιβολή τους. Ο νόμος αναφέρει ότι ουδής κάτω των 18 μπορεί να ε, παντρευτεί με ή χωρίς ε, την ε, οικογενειακή συνένεση. Έθελα να ολοκληρώσω με κάποιες ιδέες σχετικά με το τι μπορείτε να πράξετε εσείς ως Ευρωβουλευτές για να προλάβετε τους γάμους ανηλίκων. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει, πρέπει να υπάρξει στήριξη της εκπαίδευσης διότι εδώ να παραμένουν τα κορίτσια στο σχολείο είναι ένα εμπόδιο για να τις ε, μπαδεύσουν. Δεύτερον, μπορείτε Έχω δύο ακόμα σημεία και θα τελειώσω. Το θέμα της οικονομικής ενδυνάμωσης ε, των κοριτσιών θα μπορούν, να μπορούν να βρουν δουλειά όταν τελειώσουν τις, ε, το σχολείο ή τις σπουδέ τους. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, έχει καθυστερήσει στον πρόθεση ενός προγράμματος και θα πρέπει να δουν τα αποτελέσματα αυτής της εκστρατεία στο μέλλον θα πρέπει να ανανεωθούν. Συγγνώμη, αλλά το χρόνος είναι πρόβλημα στο Κοινοβούλιο. Μου είπαν ότι ε, θα έχω 15 λεπτά. Ο χρόνος κοστίζει. Λυπάμαι, πρέπει να διακόψετε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας είπατε για την εργασία που προωθεί το Plan International. Είναι πολύ σημαντική η μελέτη σας, η έκθεση. Είναι διαθέσιμη σε όλους μας. Κύριε Γκούσταψον, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά, αν δεν καταλαβαίνετε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο αλλά και την ομιλήτρια για την παρουσίασή της. Το θέμα το οποίο θίξατε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι κρίσιμη σημασία να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί χωρίς ε, ισότητα μεταξύ των φίλων ποτέ θα καταφέρουμε να έχουμε καλή ανάπτυξη και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Γιατί ε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα ο γάμος ανελίκων σε αυτές τις χώρες. Η εκπαίδευση λοιπόν για τα κορίτσια συνδέεται πολύ στενά με την καταπολέμηση του γάμου των ανελίκων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερως για το έργο σας. Τώρα, ένα ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι το εξής. Αρχίσατε την παρουσίασή σας και δυστυχώς δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε. Και περιγράψατε τα όσα θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, μας δώσατε τα μισά από τα όσα θέλατε να μας πείτε. Ίσως όμως μπορείτε να μας ε, πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα τι λείπει, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα σε αυτό το τομέα. Με συγκεκριμένους όρους τώρα, επειδή ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα υπάρχουν ε, κάποιοι απτοί στόχοι τους οποίους ε, πρέπει να επιδιώξουμε. Πρέπει να έχουμε κάποιους ε, δείκτες. Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα κατά τη γνώμη σας. Ο κύριος Φένσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ομιλητήρια για την παρουσίαση. Στον Μπαγκλαντές από το 1929 είπατε ότι ισχύει νόμος που απαγορεύει τον γάμο ανηλίκων και νομίζω ότι πρέπει να διαρωτηθούμε πώς μπορεί, μπορούμε να επερασπιστούμε τον νόμο αυτόν και να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Να παρέχουμε δηλαδή αναπτυξιακή βοήθεια στον Παγκλαντές. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν ε, όροι στην αντοξιακή βοήθεια που δίνουμε. Ιδίως όταν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους ε, φαινόμενα, όπως ε, ο γάμος των υλικών. Να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή για δύο λεπτά και μετά για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μαξάν Στοβλά από την Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την δυνατότητα να εκφέρουμε άποψη του ζητήματο. Ευχαριστούμε και για την παρουσία παρουσίαση. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι βεβαίω δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε καλύψει αυτό το θέμα με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμοστεί από κοινού με τη UNICEF στην περίοδο 2009-2012 για την καταπολέμηση του πρόωρου γάμου αλλά και κατά, της, ε, κατά το ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων. Και τέσσερα κράτη υιοθέτησαν ειδικού ε, νόμους ε, για την απαγόρευση αυτής της πρακτικής. Έχουμε μια γενικότερη προσέγγιση για την προστασία των ε, δικαιωμάτων του παιδιού και πιο συγκεκριμένα για τον γάμων υλίκων. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της δράσης μας για την καταπολέμηση παραδοσιακών πρακτικών που θεωρούμε ότι βλάπτουν τα παιδιά. Όπως ανέφερα προηγουμένως ο κατηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, ε, βία κατά των ε, παιδιών στις κοινότητες και στα σχολεία. Είναι μια διάσταση λοιπόν που έχουμε ε, υλοποιήσει πλήρως και εντάσσεται και στην επόμενη στρατηγική μας 2014-2020 αλλά και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνδέεται και με την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. αλλά και στο πρόγραμμα για τις ε, ε, παγκόσμιες προκλήσεις, ε, όπου έχουμε και εστιασμένες δράσεις για την ευμερία των παιδιών. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι έχουμε στρατηγικές που ακόμα και αν δεν έχουν άμεσο στόχο την καταπολέμηση των πρακτικών, έχουν αυτό τον αντίκτυπο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των κοριτσιών, την καταγραφή των γεννήσεων, γιατί και αυτό ε, συμβάλλει, έχει τον, ε, τη συμβολή του και τη σημασία του και πρόσφατα έχουμε και ε, πρόσκληση υποβολή ενδιαφέροντος για ένα project για τις εγκυμοσύνες κατά την εφηβεία αλλά και θέλουμε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική καταπολέμηση, καταπολέμησης αυτής της πρακτικής που συνδέεται με τον γάμο ανηλίκων. Τρέχει το, αυτή η πρόσκληση πολύ ενδιαφέροντο μέχρι τα τέλη του έτους. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ε, έχουμε και μία εργαλειοθήκη για την συστηματική ένταξη των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες ε, τις ε, δράσεις σε προγράμματα, project, πολιτικά διαβήματα. Μόλις έχει δημοσιευθεί χάρη στην UNICEF, επομένως θα τη διανύμουμε. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Εξωτερική Υπηρεσία Δράσης, κύριος Ματέο Γκομεράτο. Για δύο λεπτά. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρονικό περιθώριο που σας δίνετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ ε, το Τμήμα Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων. Δυστυχώς ε, δεν είναι εδώ ο εκπρόσωπος ε, αρμόδιες ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως έχω κάποιες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω εξ ονοματός του. Τώρα, να σχολιάσω όσα είπε ο συνάδελφος από την Επιτροπή, μέσω συστηματικής ε, και συνεχιζόμενη δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεχώ απευθύνει εκκλήσει για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και στο πλαίσιο τη εξωτερική μα δράση. 60 ε, αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο έχει θέσει προτεραιότητα τα δικαιώματα του παιδιού στι ε, στρατηγικέ Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θίγουμε συστηματικά και στους διαλόγους μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και την ενδυνάμωση των ε, γυναικών καθώς και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το στρατηγικό σχέδιο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έχουν θέσει προτεραιότητα και δράσεις που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των πρόωρων και βεβαιασμένων γάμων που πλήττουν ανηλίκους. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αυτή τη στιγμή μαζί με το Βέλγιο προετοιμάζει ε, σχέδιο όρων αναφοράς για μια διπλωματική εκστρατεία που έχει ως στόχο ε, να προσελκύσει περαιτέρω πολιτική στήριξη για την καταπολέμηση των πρόωρων και βεβαιασμένων γάμων ανηλίκων και να προωθήσουν τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών σε όλο τον κόσμο και οικονομική στήριξη παρέχεται, όπως ε, τόνισε και η Επιτροπή, μέσω της Ευρωπαϊκής ε, Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πέραν ε, των διμερών πρωτοβουλειών υπάρχουν πρωτοβουλίες και σε πολύπλευρο, πολυμερές επίπεδο. Υπάρχει η εκστρατεία ε, καταπολέμησης των πρόωρων και βιβιασμένων γάμων ανηλίκων που κερδίζει σε δυναμική τελευταία Και το 2013 είχαμε αντίστοιχη πρωτοβουλία για την κατάσταση των γυναικών που έχει αυξήσει τη δέσμευση για την καταπολέμηση ε, της ε, βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Δίνεται ιδιαίτερη εστίαση πλέον στην πρόληψη. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Τανιά Κόξ για τρία λεπτά για να απαντήσει ε, στις ερωτήσεις. Τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε γραμμές προπολογισμού για τα παιδιά, για να ε, εντοπίζουμε ακριβώς πώς ενταπανώνται αυτά τα κονδύλια. Μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και σίγουρα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ε, τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων ε, δικαιωμάτων του παιδιού. Για παράδειγμα και το σχέδιο δράση τη εξωτερική υπηρεσία δράση θα μπορούσε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη σφαιρική τέτοια προσέγγιση για τους όρους, την αρισιμότητα που συνδέεται με τη στήριξη. Εγώ δεν είμαι κατά, όμως θα πρέπει να ε, συνδέεται με τις πραγματικά πολύ σημαντικές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι δηλαδή εκεί στις χώρες όπου θα έπρεπε κάποιες χώρες να κάνουν κάτι παραπάνω, αλλά υπάρχουν κάποιοι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι ε, που δεν το κάνουν. Ή όταν υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους και δεν έχουν καλύτερες επιλογές. Εδώ, για παράδειγμα, υπάρχει ο ρόλο ε, τη ε, κοινωνικής προστασίας. Αν το κράτος μπορεί να παρέχει κοινωνική προστασία, τότε σίγουρα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό ε, στο να κρατήσουμε και τα παιδιά μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε κονδύλια, πολύ συχνά είναι περιορισμένα. Και ένα από τους λόγους είναι επειδή, για παράδειγμα, οι επιχειρήσει δεν καταβάλουν φόρους στις χώρες όπου ενεργοποιούνται, δραστηριοποιούνται. Επομένω, οι ευρωπαϊκέ εταιρείε θα μπορούσαν να καταβάλουν φόρου στι χώρε όπου δραστηριοποιούνται και να αφήσουν έτσι και τον ε, προπολογισμό αυτών των χωρών. Πολλέ από αυτέ τι χώρε δεν θα ήταν τόσο φτωχέ αν ε, γινόταν αυτό. Αν δεν ήταν φορολογική παράδεση δηλαδή. Εσεί, οι ευρωβουλευτέ, όταν ε, επισκέπτεστε αυτέ τι χώρε εταίρου, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν εκεί στους ομοτήμους σας ή ε, άλλους αξιωματούχους ε, θίγατε τη σημασία της ε, ποιοτική νομοθεσίας για την καταπολέμηση και την απαγόρευση της, των γάμων ανηλίκων, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των κοριτσιών και βεβαίως να ενισχυθούν μέτρα για την εκπαίδευση και τις καταχώρηση γεννήσεων ή τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχουν τέτοια ζήματα, μπορείτε σίγουρα να βελτιώσετε. Ευχαριστώ. So, ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε προσωπικώς αλλά και ως πλάνο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η μερίσια διάταξη προβλέπει την παρουσίαση μελέτης για τη στρατηγική της Ένωσης στον Ειρηνικό για την ανάπτυξη. Και δίνω το λόγο στους ε, συντάκτες εκθέσεως για να μας παρουσιάσουν τα κύρια συμπεράσματα Ευχαριστώ τα στρατιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Consortium για τις ε, μελέτες στον Ειρηνικό που έκαναν τον κόπο να έρθουν μέχρι εδώ για να μας παρουσιάσουν την έκθεση και δίνω το λόγο στον καθηγητή Edvai Bidding από το Παρεπιστήμιο του Μπάριγκεν της Νορβηγίας. Έχετε τρία λεπτά όπως πάντα. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά. Για δέκα λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα PowerPoint που έχουμε ετοιμάσει. Και αν μου επιτρέπετε θέλω να το παρουσιάσω. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω για τη μελέτη αυτή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην ε, Μεσόγειο σκοπεύω να αναλύσω, να παρουσιάσω την ανάλυση και τα πορίσματα εν γέννη της εκθέσεως και μετά δώσω το λόγο στον κύριο Κρούκ, αν μου επιτρέπετε, για να, κάνω την, για να κάνει την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Έχουμε μια σειρά από συνεργάτες, ε, εκτός από τον κύριο Κρούκ και τον υποφαινόμενο. Έχουμε άλλους δύο που είναι και εδώ σήμερα παρόντες. Και Περιμένω να δω να βγαίνει στην οθόνη η παρουσίασή μου με τις διαφάνειες, όσον υπο Η περιοχή λοιπόν του Ειρηνικού, των νήσων του Ειρηνικού που θα δούμε ευθύς αμέσως στην παρουσίαση με διαφάνειες Καλά, ας συνεχίσω λοιπόν. Οι νήσοι λοιπόν του, Ατλαντι... του Ειρηνικού έχουν περίπου 12 εκατομμύρια κατοίκους από τις ε, χαμηλού ε, υψομέτρου ατόλες μέχρι τα ηφαιστειογενή εδάφη και τη Νέα Γουινέα. Άλλα θέσεις θα μπορούσαμε να περάσουμε στη δεύτερη διαφάνεια του μεταξύ. And the next one, please here we are. And I'll continue to advise on when to proceed. Uh, the biological... Η βιοπικιλότητα λοιπόν του ειρηνικού είναι παρά, βαίνει παράλληλα και με την πολιτιστική. Έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό των γλωσσών όλου του κόσμου που εκπροσωπείται εκεί και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη γραμμή της υποστήριξη της ε, πολιτιστικής ε, ποικιλομορφίας σε κάθε της έκφανση. Έχουμε λοιπόν τον μεγάλο ωκεανό, όπως λέγεται, με περιοχές απομονωμένων νησί, νησών ή αρχιπελάγων συχνά, που όμως έχει και κοινή ιστορία και εμπόριο και παρελθόν κοινό, όπως έχει χαρακτηριστεί από ένα μεγάλο ερευνητή, πρόκειται για μια θάλασσα νησιών. Υπάρχουν ε, ε, μεγάλα κράτη με 7,5 εκατομμύρια όπως Παππούα Νέα Γουινέα και πολύ μικρά μέχρι 2.000 κατοίκους. Είναι πολύ μεγάλες οι αποκλήσεις λοιπόν. Το Τουβαλού, αυτή η μικρή ατόλη, έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη με 750 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα τρίτο περίπου της αντίστοιχης ζώνης της Παπουάς Νέας Γουινέας. και σε άλλη περίπτωση έχουμε να κάνουμε τη 12η μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη και βέβαια ένα τεράστιο ποσοστό των παγκόσμιων θαλασσίων πόρων. Οι νησιώτες αυτοί λοιπόν την θάλασσα την έχουν αξιοποιήσει για τα ταξίδια και τις συναλλαγές αλλά και τις ανταλλαγές. Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια έγινε η εξερεύνηση με τα κανό του ειρηνικού. Τώρα τα πλοία χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές για την αλληλεία, κυρίως του τόνου, και έχει κέρια σημασία η θάλασσα για τις χώρες αυτές, για τα νησιά αυτά. Όμως και η στεριά δεν θεωρείται αποκομμένη από τη θάλασσα. Έχουμε οικισμούς σε ορισμένες πολύ στενές ατόλες, με πολύ, ε, πολύ εκτεθειμένους στην άνοδο του επίπεδου της θάλασσας και άλλους περιβαλλοντικού κινδύνους, που μπορεί να έχουν να κάνουν με την ξύλευση, παραδείγματι, ή την εξόριξη σημαντικών υπόγειων πόρων. Η πρόσβαση λοιπόν τόσο στη θεριά όσο και στη θάλασσα ανήκει στους κατοίκους των περιοχών αυτών με οικονομίες της υπαίθρου που ε, μετατρέπονται σιγά σιγά σε όλο και πιο εξαρτώμενες από την παγκόσμια οικονομία έχουμε να κάνουμε με πόρους τεράστιας σημασίας, είτε πρόκειται για την αλία είτε πρόκειται για την ξυλία. Στο δυτικό ειρηνικό έχουμε σχεδόν εξάντληση των ε, ε, πόρων ξυλίας και αντίστοιχα μεγάλη μείωση των αποθεμάτων των αλληλευτικών. Ε, είναι εκτεθειμένες οι περιοχές αυτές στις φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι, παλαιριακά κύματα, αλλά και η κλιματική αλλαγή τώρα, εξαρτώνται και παρουσιάζουν πολύ σημαντικά πλημμύρες, όπως την προηγούμενη εβδομάδα τη χειρότερη στην ιστορία τους έζησαν τα νησιά του Σολομώντα. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια δέσμευση στην υπόθεση αυτή. Με ένα πολύ μεγάλο λοιπόν αριθμό κρατών, με σχετικά μικρό πληθυσμό συνολικά, παραμένει εξαρτημένη από την ε, παγκόσμια βοήθεια, διεθνή βοήθεια, η περιοχή αυτή του Ειρηνικού, με τη μεγαλύτερη εξάρτηση κατά κεφαλήν. Πενταπλάσια κατά κεφαλήν από ό,τι η υποσαχάρη Αφρική για όλες τις περιοχές του Ειρηνικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη θέση στο χώρο αυτόν με το δέκατο αναπτυξιακό πρόγραμμα που προσέφερε τα τελευταία πενταετία 400 εκατομμύρια στις χώρες ΑΚΕ που ανήκουν στη ζώνη αυτή και και όλο και ενισχυόμενη γεωπολιτική ε, αντιπαράθεση των διεθνών δυνάμεων όπως η Κίνα στη ζώνη αυτή που εμφανίζεται όλο και πιο δυναμικά. Βέβαια η Γαλλία με την Νέα Καλλιδονία έχει πολύ σημαντικό ρόλο ακόμη. Οι χώρες του ειρηνικού δεν είναι παθητικοί αποδέκτες βοήθειας αλλά προσφέρουν ανταπόκριση μέσω του διαλόγου, την απορρόφηση, την αξιοποίηση της βοήθειας που τους προσφέρεται επί τόπου και παραλαμβάνουμε είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που τους προσφερθεί στον τομέα αυτόν. Και αν μου επιτρέπετε να το λέγω, στον Τόνι Κρουκ. Έχουμε να κάνουμε μια μακρά ιστορία επί, επαφής των πολιτών των κρατών αυτών με τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, συναλλαγές και ανταλλαγές με σημαντικό οικονομικό συμφέρον. Έχουμε να κάνουμε και με πολύ μεγάλη σημασία τουριστική, αλλά και με οικονομικούς φόρους όπου αναπτύσσεται ένα περιβάλλον στο οποίο η τοπική διάσταση έχει την προτεραιότητα εν τέλει. η επίτευξη ανάπτυξης, από, ε, ανάπτυξης άνωθεν που συναντά όμως και την βάση ε, κάποια στιγμή είναι μια πολύ επιτυχημένη επιλογή εταιρικής σχέσης μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Έχουμε όλο και, όλο και πιο δυνατές φωνές που ζητούν την αναπτυξιακή βοήθεια χωρίς να παίρνουν ακραία μορφή διαφορετικές μορφές όμως και ποικιλία ε, επιδιωκόμενου αποτελέσματος. παραδείγματι υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση χωρίς εξαρτήσεις, ισότιμες εταιρικές σχέσεις και περισσότερη ε, επιλογή, δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προγραμμάτων. Αυτή η κριτική μπορεί να είναι ε, πολύ σχηδής. Μπορεί η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία να είναι μέλη και κύριοι χορηγοί του σχετικού φόρουμ και να προσδιορίζουν το τι συμβαίνει μέσα από μια υπερεθνική και υπερφυσική υπηρεσία. Πάντως βλέπουμε ότι ένας υπουργός από τα κρατευτά δηλώνει ότι αν θέλει κάτι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει μέσα από την ε, Ένωση αυτής της συνεργασίας. Οι χώρες του ειρηνικού θέλουν να αναβαθμίσουν το χώρο που τους ανήκει, το χώρο που διεκδικούν μέσα στην ε, ομάδα των ΑΚΕ, αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σχέση η οποία έχει ιστορικούς ε, δεσμούς, ιστορική βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την οποία χρειάζεται να αξιολογήσουμε τις προοπτικές από την πλευρά των ΑΚΕ και το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει στο μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε στη στρατηγική για το 2020. Τέλος, θα πρέπει να δούμε, δούμε τους τρόπους με τους οποίους χρηματοδοτούν τα προγράμματα. Γενικά, η γραφειοκρατία και η διάδραση που υπάρχει αποκαλύπτουν τις προθέσεις των εταίρων. Ορισμένες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο αλλά και αρπισοπίες των Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επηρεάζονται από άμεσες ε, από τα αποτελέσματα των ε, πληρωμών και υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης. Υπάρχει ένα διάγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει για τον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ο χρόνος σας έληξε εδώ και 45 δευτερόλεπτα και μια που διαβάζετε το κείμενο όλοι μπορούμε να το αναγνώσουμε στο σπίτι μας. Το λόγο έχει ο επόμενο αγορητή. Παρακαλώ, έχετε πέντε λεπτά. Δώστε μα ε, τα βασικά μηνύματα. Πέντε λεπτά είναι πολύς χρόνος για να μας πείτε μερικά πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δράτω με τις ευκαιρία ε, να ευχαριστήσω την ΕΚΟΠΑΣ για την δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας ε, για αυτή την παρουσίαση της έκθεσης ονομάζομαι Ιδρυκτεύη και δουλεύω για την Διεθνή Οργάνωση για την διατήρηση της ε, βιοποικιλότητας. Θα ήθελα να μιλήσω για το περιεχόμενο της έκθεσης και αγαπητή Πρόεδρε μέλη του Κοινοβουλίου θα αναφέρω τρία, τρία θέματα που μας απασχολούν. Όπως είπαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής στον Ειρηνικό ωκεανό, στον του Ειρηνικού και οι ε, προτεραιότητες ε, έχουν διαπιστωθεί από την EDF και το Ταμείο αναπτυξιακής βοήθειας. Θα ήθελα να προτείνω και να καλέσω τα μέλη του Κοινοβουλίου να λάβουν υπόψη τους ότι σε πολλές περιπτώσεις στο ειρηνικό υπάρχουν χρηματοδοτήσεις οι οποίες βασίζονται σε προγράμματα αλλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντα στις στρατηγικές που έχουμε προωθήσει σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να προτείνουμε πως χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων στον ειρηνικό. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα, θα πρέπει δεν θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φυσικά τα προγράμματα σας είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προγράμματα αφορούν μία πτυχή και δεν ε, είναι έχουν συλληφθεί με βάση ε, μιας, ολοκληρωμένου προγράμματος. Τώρα, σε ό,τι φορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής τους, έχετε ήδη υπογράψει 35 δισεκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση. Το μίσο όμως θα ήθελα να προτείνω να εστιάσουν τα χρηματοδοτήσει της ε, Ένωσης είναι οι τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη επαρκώς από τα υπόλοιπα προγράμματα και αφορά την ε, ζήτημα της αποκατάστασης ε, για λόγους ανάπτυξης. Πολλές φορές αυτό δεν καλύπτεται από την ε, βοήθεια που παρέχουν τα ταμεία συχνά οι απαντήσεις ε, αφορούν κατα... καταστάσεις και δεν προβλέπουν αποκατάσταση. Προτείνω λοιπόν, Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, ότι η συμμορδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εστιάσει στο μέλλον σε αυτά τα θέματα σε ό,τι φορά τις αλλαγές του κλίματος. Το τρίτο σημείο, Πρόεδρε, είναι το δυναμικό για συνεργασία γύρω από τα θέματα τεχνολογίας των ενώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα μια εστίαση σε τεχνολογία η οποία καθοδηγείται από την έρευνα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ότι οπουδήποτε αλλού και μιλάω για την αϊφόρο θαλάσσια μεταφορά Μιλάμε για την χρησιμοποίηση του αέρα των ανέμων και την εκμετάλλευσή του. Είδαμε εικόνες ε, από κανό τα οποία ε, ε, τον ειρηνικό και την τεχνολογία αυτή την χάσαμε, την απολέσαμε. Όμω εσεί στην Ευρώπη συνεχίζετε να έχετε αυτή την τεχνολογία. Αυτό που θα θέλαμε να προτείνουμε λοιπόν είναι να υπάρξει μια κάποια ανταλλαγή απόψεων γύρω από την αιωλική ενέργεια και το πώς θα αναπτύξουμε τους τρόπους μεταφοράς χρησιμοποιώντα την αιωλική ενέργεια. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κέβιν και για το ότι τηρήσατε το χρόνο σας. Ο κύριος Πόγκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συντάκτες της μελέτης, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ως Ευρωβουλευτής προέρχομαι από την περιοχή του Ειρηνικού, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η περιοχή αυτή ε, εξετάζεται σήμερα από πλευρά ε, της Επιτροπής μας και η μελέτη καταδεικνύει την γεωστρατηγική σημασία αυτής της ε, περιοχής του Ειρηνικού λέγεται ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα αφορούν τον άξονα Ασία ειρηνικό. Είναι λοιπόν πολύ καλό το ότι η Κομισιόν εξετάζει το ζήτημα. Συμφωνώ με την μελέτη για την ύπαρξη μιας πραγματικής συντατική σχέσης και να απομακρυνθούμε από την ε, ε, σχέση ε, δωρητή και δικαιούχου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένα σωστό συντονισμό της βοήθεια, το οποίο θεωρώ απαραίτητο. θέσω μία απλή ερώτηση στους συντάκτες της μελέτης, δηλαδή πώς θα μπορούσε να γίνει να χρησιμοποιήσουμε τις υπερπόντιες ε, περιοχές που βρίσκονται στην περιοχή αυτή του ειρηνικού έτσι ώστε να καταστούν πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περιοχή του Ειρηνικού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υπερπόνη διαμερίσματα ως πρέσβεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νόησερ, έχετε το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς εκείνους οι οποίοι κατήρθησαν και παρουσίασαν αυτές τις εκθέσεις. Αναφέρθηκαν σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τομείς όπου όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει πιο ενεργή δράση. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία στην αναπτυξιακή πολιτική κοινή μαζί και με άλλους χορηγούς όπως η Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Θα ήταν πολύ σημαντικό, παραδείγματι, εδώ, αν μπορούσαμε να επεξεργαστούμε μια κοινή στρατηγική, ώστε να βοηθήσουμε καλύτερα, όπως μπορούμε, τα κράτη αυτά του ειρηνικού. Ο δεύτερος τομέας που δεν εξετέθη τόσο πολύ ήταν, ε, αλλά αφορά εμάς ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτός των ε, φορολογικών παραδείσων που εδρεύουν στον ειρηνικό. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και όταν προσπαθούμε να ε, περιορίσουμε, να εξωτερώσουμε τους φορολογικούς παραδείσους από τον κόσμο, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των φορολογικών παραδείσων στον ειρηνικό. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό του, ε, των φυσικών πόρων, των υπόγειων κυρίως ορυκτού πλούτου κτλ. που έχουν τα κράτη αυτά και που βεβαίως ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα βιομηχανικά κράτη. Μόνο στο κοινό εμπόριο μπορούν τα κράτη αυτά του ειρηνικού να διαχειριστούν αυτόν τον πλούτο. Με κοινή διαχείριση δηλαδή. Με κοινή διαχείριση επίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ένα άλλο θέμα, γιατί με λύπη βλέπω ότι υπάρχει μόνο μία μεμονωμένη αλληλευτική συμφωνία με το Κυριμπάτι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κυριμπάτι λοιπόν, ένα νησιωτικό κράτος και ενώ όλα τα υπόλοιπα θέλουν να έχουν μια διαφορετική στάση, εξαγοράστηκε, θα το πω κάπως σκληρά, και προχώρησε στην σύναψη αυτής της ελευθερικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και με τέτοιου είδους συμφωνίες να ε, χειριζόμαστε τα θέματα συνολικά σε συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα λάβω και εγώ το λόγο, λέει η Πρόεδρος, για μια ερώτηση. Θέλω να μάθω εάν το Πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό σας τούτο έχει προβεί σε συνολική αξιολόγηση των αλληλευτικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Ειρηνικού σε σχέση με τους αλληλευτικούς σπόρους και τις συνέπειες σε αυτούς. Και θέλω να ρωτήσω εάν φρονείτε ότι ο σημαντικότερος αλληλευτικός σπόρος, ο τόνος δηλαδή, ε, την χάνει καλής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή, μάλλον Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με την κυρία Κάρμεν Ρούις Σαράμου. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Είμαι Κάρμεν Ρουής, επικεφαλής ε, του τμήματος ε, για τον Ειρηνικό στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πολύ σύντομα. Με συνοδεύουν δύο συνάδελφοι δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Χαιρετίζουμε ε, την μελέτη για την περιοχή του Ειρηνικού που δυστυχώς ως ε, περιφέρεια δεν βρίσκεται στο προσκήνιο επίπεδο κάθε μέρα. Επομένω, έστω και για μισή ώρα χαιρόμαστε που συμβαίνει αυτό που είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε αυτή τη παρουσίαση της μελέτης από το ΕΚΟΠΑΣ. Για εμάς, ε, στην υπηρεσία εξωτερική δράση, το πιο σημαντικό είναι η σφαιρική πολιτική συνοχή σε αυτή την περιφέρεια. Πολλοί είναι οι φορείς ε, και οι παράγοντες που δρούν εκεί και δεν μιλώ μόνο για δωρητές, υπάρχουν και άλλες ε, ε, κλαδικές πολιτικές ε, για τον ειρηνικό, αναφέρουμε για παράδειγμα στην αλληλεία, για το εμπόριο, ε, με διάφορες επιμέρους εμπορικές διαπραγματεύσεις. Και εμείς με, από τη μεριά μας προσπαθούμε να συνδιαλλαγούμε με όλους αυτούς ε, τους ε, φορείς ε, για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, πληροφορίες, τη γνώση μας για όλες αυτές τις πολιτικές στην περιφέρεια του Ειρηνικού και για να έχουμε την καλύτερη δυνατή πολιτική συνοχή. Γιατί διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε μόνο κακές πολιτικές. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, θέλουμε να πάμε παραπέρα Πέρα λοιπόν από αυτές τις παραδοσιακές ε, σχέσεις και εταιρικέ σχέσεις που ε, βασίζονται περισσότερο σε σχέσεις ε, δωρεάς, του δωρητή δηλαδή και του παραλήπτη της δωρεάς. Και εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο με καθένα από τα 15 κράτη-μέλη της περιφέρειας Ειρηνικού για να συζητήσουμε κοινέ αρχές, κοινέ αξίες πέραν της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αναφερόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διάσταση του φύλου που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην περιφέρεια του ελληνικού και προηγουμένως ακούσαμε ε, και το προηγούμενο θέμα για το γάμο ανηλίκων. Προσπαθούμε λοιπόν να πάμε πέρα από τα μόνιμα σημεία στην ημερήσια διάταξη που μέχρι τώρα ήταν η ανάπτυξη και το εμπόριο. Υπάρχουν πολλές, πολλοί στόχοι σε ό,τι φορά τις κοινέ αξίες που μπορούμε να έχουμε με τον ειρηνικό. Και τέλος, η περιφέρεια του ειρηνικού είναι ιδιαίτερα μεγάλη, περίπλοκη και ετερογενής, όπως ανέφεραν και οι πρόσωποι του ΕΚΟΠΑΣ. Επομένως, αναπτύσσονται και πολλές ε, περιφερειακές δομές ή υποπεριφερειακές δομές. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως είναι το φόρουμ ε, νήσων του Ειρηνικού, που λειτουργεί με πολιτικό γνώμονα, αλλά και με συμμετοχή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Πολλά, λοιπόν, πολλές λοιπόν είναι οι θετικές εξελίξεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόμαστε με το καλύτερο τρόπο. Δηλαδή ότι το καλύτερο είναι να το αναλάβουν μόνοι τους. Εμείς ε, έχουμε να κάνουμε μια περίπλοκη κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο που θα επιλέξουν οι ίδιες οι χώρες ε, του ειρηνικού. Δεν ξέρω αν έχω κι άλλο χρόνο. Όχι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Merci de vos Ευχαριστώ που πήρατε και αυτό το ζήτημα υπόψη, το θέμα του χρόνου. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα το λόγο στο consortium για να απαντήσει. Έχετε πέντε λεπτά να μοιραστείτε και οι τρεις σας. Πώς θα γίνει αυτό, θα το επιλέξετε εσείς. Ξεκινάμε λοιπόν με το καθηγητή Βιντίνγκ, που πήρε πρώτος το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω εν συντομία στο ζήτημα της αλίας που εφήγει στο τέλος. Ήθελα να πω ότι στον ειρηνικό υπάρχουν πολλά έθνη που εκφράζουν ε, την κυριαρχία τους κυρίως μέσω της αποκλειστικής ε, οικονομικής ζώνης, όχι μέσω της ταιριάς που είναι πολύ μικρή ως ε, επιφάνεια. Γι' αυτό τα ζήτημα που αφορούσαν τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυριμπάση είναι αξιοσημείωτα γιατί αναπτύσσουν ακριβώς αυτές τις ιδέες ε, τη αυτοκυριαρχία, Όμως, της εθνική κυριαρχίας. Όμως, αν λάβουμε υπόψη και τον ιδιαίτερα καινοτόμο ρόλο των ε, περιφερειακών συστημάτων διαχείριση της αλίας, που ε, ελέγχουν για δεκαετίες τα δύο τρίτα των αποθεμάτων ε, τόνου, θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη όταν εξετάζουμε τους αλευτικούς πόρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Διάσταση του φύλου πρέπει να αναγνωρίσουμε το περιορισμένο πεδίο εφαρμογή που έχουμε με μια τέτοια μελέτη, αλλά και να πούμε ότι ε, μέσα στη σύμπραξή μα υπάρχουν ε, και άλλε διαργασίε. Είχαμε πέρυσι ένα εργαστήρι για τη ε, διάσταση του φύλου και τη βία κατά των γυναικών αλλά υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση. Συνεργαζόμαστε με την ΤΕΦΚΟ για να έχουμε ένα ευρύ ε, project που να αφορά ε, τις γυναίκες. Υπάρχει διαφοροποίηση ό,τι αφορά και ε, τα πολιτικά μορφώματα και τα OCTs είναι πολύ σημαντικό τμήμα της συμβολής μας. Επομένω, η περαιτέρω ολοκλήρωση του OCT είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο ε, συστήνει η μελέτη είναι η αναθεώρηση της επισκόπησης που είχε γίνει για μελέτη σκοπιμότητας σε συγκεκριμένα θέματα. Να τα εντάξουμε όλα αυτά στο ίδιο πλαίσιο και να έχουμε περισσότερες άμεσες επαφές ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή. Και έτσι σίγουρα και οι OCT θα μπορούν να έχουν αυτό το ρόλο πρεσβευτού. Τώρα, για την εξόριξη στον πυθμένα της θάλασσας είναι κάτι το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα και η Παππού Ανέγου η Νέα είναι η χώρα που περιμένουμε να ανταποκριθεί ε, πρώτη. Αλλά αυτό αφορά και τον ρόλο με τον οποίο μεταβάλλεται η ε, περιοχή. Η Παππού Ανέγου η Νέα λοιπόν γίνεται ένας ε, περιφερειακός φορέας ε, αλλαγής. Κατά τη γνώμη μου θα αναπτύξει αυτή την ε, εμπορική δραστηριότητα η Παπώνε Γουινέα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Ε, συνεχίζω για την περιοχή του Ειρηνικού αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της πρόληψης προς ε, την εξόριξη στο βυθμένα της θάλασσας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πόροι, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όταν αν και όταν ε, προβούμε σε τέτοια εξόριξη, δεν θα γίνει αυτό σε βάρος ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε προς τους εταίρους μας. Για τα OCTs και την συμμετοχή τους στις εταιρικές σχέσεις στον Ειρηνικό. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο Πόγκα, τον κύριο Ευρωβουλευτή που έθιξε αυτό το ζήτημα. Βεβαίω ε, και η Νέα Καλλιδονία τώρα ε, βρίσκεται επικεφαλή τη αρμόδια ομάδα. Ω λοιπόν υποπεριφερειακό μόρφωμα, το OCT ήδη συμμετέχει και ηγείται ενό από αυτούς τους υποπεριφερειακούς φορείς που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην περιοχή. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν κυρία Πρόεδρε ήδη έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Για την αλληλεία μπορώ μόνο να επιστρέψω το ερώτημα στα επόμενα 15 δευτερόλεπτα. Γιατί έρχεστε στον ειρηνικό, γιατί ακριβώς έχουμε τα αποθέματα του τόνου. Και αν τα έχουμε τα αποθέματα τόνου, είναι δικά μας τα αποθέματα. Και αφόσον πρόκειται για δικά μας αποθέματα, εμείς πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε πότε, πώς και σε ποια τιμή θα σας τα πουλήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μένει μόνο να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρουσιάσεις, την παρουσίαση αυτής της μελέτης που θα είναι πολύ χρήσιμη για τις μελλοντικές μας εργασίες. Τώρα μπορούμε να περάσουμε σε μια επόμενη μελέτη για τη δυναμική της ε, κοινωνικής ε, οικονομίας για την ε, τοπική ανάπτυξη στην Αφρική. Αυτή η μελέτη εκπονήθηκε από το Έλισις. Να ευχαριστήσω την κυρία Τζούλια Γκαλέρα που είναι εδώ μαζί μας για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Έχετε το λόγο κύρια Γκαλέρα. Για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσετε τη μελέτη σας. Thank you, Madam Chair, for me the floor. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που δίνετε τον λόγο. Ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και, και τους διάφορους εκπροσώπους για τη συμμετοχή του σήμερα. Όπως αναφέρει και ο τίτλος της μελέτης, θα παρουσιάσονται κύριε ευρήματα μιας ε, ερευνητικής ανάλυσης ε, των δυνατοτήτων ε, της κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη της Αφρικής. Πολλά πρέπει να, ακόμα να γίνουν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση τη κατάσταση κοινωνική οικονομία στην Αφρική. Παρ' όλα αυτά, η αναθεώρηση τη υφιστάμενη ε, βιβλιογραφία ε, και τη κατάσταση σε τέσσερι χώρε, Γκάν, Αιθιοπία, Μαρόκο και ε, Κένια, μα επιτρέπει να τλήσουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα και να καταλήξουμε σε κάποιε αρχικέ συστάσει. Οι οργανώσει που ανήκουν στον χώρο τη κοινωνική οικονομία πάντα επέμειναν να δημιουργήσουμε και όχι να καλύψουμε την αξία γενικά εξαιρείται η ε, επιδίωξη του κέρδους ε, και η απόδοσή τους στους ε, ιδιοκτήτες ως στόχος. Όμως έχουμε ως στόχο την προώθηση του γενικού συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Από την νομική σκοπιά η κοινωνική οικονομία συνήθως ορίζει διάφορες, διάφορους και τέτοιους λόγους. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία της οικονομίας η κοινωνική οικονομία είναι αυξανόμενος φορέας της αφρικανικής οικονομίας, όμως δεν αναγνωρίζεται αντιστοίχω. Ο όρος κοινωνική οικονομία δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Αφρική ούτε από ε, τους υπεύθυνους για ε, τη λήψη αποφάσεων και τους ερευνητές. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική οικονομία σε αυτές τις χώρες. Αντιθέτως μπορούμε να πούμε ότι η Αφρική είναι η Ήπειρος όπου η κοινωνική οικονομία ε, διαδραματίζει τον ε, πιο ε, σημαντικό ρόλο καθώς καλύπτει μεγάλο αριθμό οργανισμών που έχουν και κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και πολλές δραστηριότητε μεταξύ άλλων και παραγωγή ε, εμπορευμάτων ε, και προϊόντων. Μπορεί βεβαίως να δημιουργήσει προβλήματα γιατί αγνοούμε τις παραδόσεις κάποιες φορές που υφίστανται σε αυτές τις χώρες και για να το αποτρέψουμε αυτό έχουμε προσαρμόσει τα όρια της κοινωνικής οικονομίας για να λαμβάνουμε υπόψη και την διάσταση της αυτοβοήθειας που υπάρχει στην Αφρική. Γι' αυτό έχουμε εντοπίσει διάφορες μορφές ε, οργανισμών. Διακόπτη η Πρόεδρος, συγγνώμη, αλλά πρέπει κάπως να μιλήσετε λίγο πιο αργά. Υπάρχει διερμηνία σε 20 χώρες, δεν πρέπει να διαβάζετε, πρέπει να μας τα λέτε. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό το κίνδυνο, έχουμε προσαρμόσει τα όρια τη κοινωνική οικονομία για να λαμβάνουμε υπόψη και την ε, παράδοση τη αυτοβοήθεια που υπάρχει ή τη αμοιβαία βοήθεια που υπάρχει στην Αφρική. Έχουμε εντοπίσει διάφορε μορφέ οργανώσεων. Συγκεκριμένα έχουμε άτυπε ομάδε αυτοβοήθεια που καλύπτουν ένα πολύ σημαντικό κενό από την έλλειψη επίσημων θεσμών. Επιπλέον, έχουμε το παράδειγμα των συνεταιρισμών. Ε, αντίθετα με την Ευρώπη, όπου ε, αποτελούσε ένα ε, άνωθεν φαινόμενο, στην Αφρική πρώτα υπήρχε από τις αφρικανικές κυβερνήσεις αυτός ο θεσμός. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποιες χώρες υπάρχει αναζωογόνηση των παραδοσιακών αυτών μοντέλων συνεταιρισμών. Τέλος, κάποιες φορές έχουμε και διάφορους λόγους με τη μορφή κάποιες φορές των ΜΚΟ που δρούν ε, γύρω από ένα συγκεκριμένο σκοπό, είτε αυτός είναι οικονομικός, κοινωνικός ή ανθρωπιστικός. Δεύτερο συμπέρασμα, η κοινωνική οικονομία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, η κοινωνική οικονομία παρέχει στις ε, τοπικές κοινότητες ε, το θεσμικό πλαίσιο για την επαρκή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πολιτών να επιλύουν ε, διάφορα κύρια ζητήματα ε, μέσω της παροχής, για παράδειγμα, ε, επιστηστικής ασφάλειας, πρόσβασης στο νερό και στην ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία και το καθεξής. Γι' αυτό ενδυναμώνουν ε, τους ε, πλέον αδυνάτους ε, και αυτό γίνεται με τους περιορισμένους πόρους που έχουν στη διαθεσή τους πολλές φορές. Ο αντίκτυπος λοιπόν αυτός μπορεί να ειδωθεί από πολλές σκοπιές, συμβάλλει στη μείωση της ένδυας και την στήριξη της βιώσιμης οικονομίας. Συμπληρώνουν λοιπόν τις υπόλοιπες δομές που υπάρχουν και παρέχουν υπηρεσίες που οι παραδοσιακές δομές δεν παρέχουν. Άλλα παραδείγματα μας δίνουν ε, διάφορες επίσημες ή αναπίσημες ε, γεωργικές δομές, στην Κάνα για παράδειγμα, που συμβάλλουν ε, σημαντικά στην αδυνάμωση των μικρών γεωργών. Αντίστοιχο παράδειγμα υπάρχει και στην Αιθιοπία, που συμβάλλει στη μείωση της ένδυας περισσότερο από ότι άλλες μορφές τέτοιων οργανώσεων. Όμως, οι οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προστασία της οικονομικής σταθερότητας. Ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ο κύριος ρόλος ε, των συνεταιρισμών ε, σε κάποιους ε, τύπους ελαίων για τη στήριξη των γυναικών που έχει βελτιώσει την θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Και έτσι μπορούν οι γυναίκε να έχουν και τη δική τους φωνή που ακούγεται στις παραδοσιακές μουσουλμανικές ε, κοινωνίε. Τέλος, ε, αυτοί οι οργανισμοί συμβάλλουν σε πιο ισορροπημένη χρήση και κατανομή των πόρων. Χάρη στη συμμετοχή των ε, τοπικών ενδιαφερμένων μερών, τέτοιε οργανώσεις ε, προωθούν ε, την συμμετοχική δημοκρατία και τις τυχές ε, δομές που συμβάλλουν σε καλύτερη λήψη αποφάσεων στο στρατηγικό επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στη δράση και την ανάπτυξη της δράσης αυτών των οργανώσεων. Κύριο εμπόδιο οφείλεται στην έλλειψη αναγνώρισης της κοινωνικής οικονομίας που πολύ συχνά οδηγεί σε ανεπαρκές νομικό πλαίσιο και αναποτελεσματικές πολιτικές. Όπως δείχνει και η ευρωπαϊκή εμπειρία, η στήριξη και, και το καλό νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικός, ε, σημαντική κινητήρια δύναμη για αυτές τις οργανώσεις. Ωστόσο, στην Αφρική οι δημόσιες πολιτικές πολύ συχνά δεν ε, παρέχουν ε, στήριξη, είτε γιατί υπάρχει ευρύτερη έλλειψη, ε, τέτοιων πολιτικών, είτε επειδή τεχνικά, τεχνητά μεταφέρονται από το δυτικό πλαίσιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ε, αυτών των χωρών. Άλλος παράγοντας ε, ενδυνάμωσης της ανάπτυξης και αντικτύπου στην κοινωνία είναι η διαθεσιμότητα αντίστοιχων δομών για αυτές τις οργανώσεις. Τα ευρήματα αυτή τη μελέτη οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ στήριξη. Πρώτον, είναι σημαντικό η κοινωνική οικονομία να αναγνωρίζεται στην Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει ε, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ύπαρξη τέτοιας κοινωνικής οικονομίας στην Αφρική και για τη στήριξή της στη μείωση της ένδυας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο ε, στην διευκρίνηση των βασικών ρόλων ε, επιμέρους ε, οργανώσεων που διαδραστηριοποιούνται στην Αφρική για να αυξηθεί η ευθυτοποίηση σε ό,τι φορά την κοινωνική οικονομία για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης οικονομίας. Και και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ό,τι αφορά τον ρόλο των ίδιων των ε, οργανώσεων σε διάφορου τομεί τη οικονομία. Μεταξύ άλλων, πρόσβαση στην ε, κοινωνική πρόνοια, επιστημική ασφάλεια, στέγαση, μεταφορέ ε, και εκπαίδευση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει στην κοινωνική οικονομία σε ευρωπαϊκές πολιτικές στήριξης, να μπει λοιπόν στον κατάλογο των άλλων μη κρατικών φορέων που αναφέρεται στο κατάλογο των εταίρων με την Αφρική. Να ενδυναμώσουμε λοιπόν και να, ενθαρρύνουμε ε, τους, ε, τις αντιπροσωπείες ε, που πηγαίνουν στην Αφρική για να προσκαλούν αυτές τις ε, οργανώσεις, τις διαβουλεύσεις. Για να κατανοήσουμε το ρόλο και τη δυναμική της κοινωνικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει και νέα νέο ερευνητικό έργο για τη χαρτογράφηση τη κοινωνική οικονομία σε όλε τι χώρε Αφρική, ε, να συλλέξουμε νέα δεδομένα που μπορούν ε, να στηρίξουν και να αποδείξουν την ε, σημασία του κλάδου και να εντοπίσουμε και καλές βέλτιστες εμπορικές πρακτικές ε, που έχουν θεσμοθετηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Μετά, τα εφιστάμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανταξιακή Συνεργασία με την Αφρική, θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση τέτοιων ε, ε, προγραμμάτων που μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες ε, αυτών των οργανώσεων στην Αφρική. Με την στήριξη και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Να διευκολύνουμε την άντληση διδαγμάτων από ομοτήμους και να δώσουμε νέες δυνατότητες σε νέα κρατημέλη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τέτοιες ε, αποτελεσματικές ε, δομές κοινωνικής οικονομίας. Να έχουμε αντίστοιχες δομές που θα στηρίζουν την ανάπτυξη και την αύξηση δυναμικού αυτών των οργανώσεων. Να έχουμε αντίστοιχη χρηματοδότηση για να βοηθούμε την σύσταση και ανάπτυξη αυτών των οργανώσεων και να ενθαρρύνουμε αντίστοιχα δίκτυα βορρά-νότου και νότου-νότου ε, για τη στήριξη αυτή τη κοινωνική οικονομία. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει συνδέσει και με άλλου διεθνεί οργανισμούς για να στηρίζει την ε, ανάπτυξη ενό ε, κατάλληλου περιβάλλοντο για τι διάφορε οντότητε που συνιστούν την κοινωνική οικονομία στην Αφρική να ενθαρρύνουμε τους Αφρικανούς υπεύθυνους λύσης πολιτικής για την θεσμοθέτηση κατάλληλου νομικού πλαισίου που επιτρέπει την αποτελεσματική δράση διαφόρων μορφών τέτοιων οργανώσεων και τον περιορισμό πορτονοστικών συμπεριφορών. Να στηρίξουμε την ε, θέσπιση ε, τοπικών εταιρικών σχέσεων που προωθούν την ανάπτυξη αυτών των οργανώσεων. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Μάλιστα, κύριε Σμίτσελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κυρία Γκαλέρα για την παρουσίασή σας. Σύντομες παρατηρήσεις. Η κοινωνική οικονομία εντοπίστε στο χώρο ανάμεσα στο δημόσιο, στο κρατικό και το ιδιωτικό πεδίο. Εμείς έχουμε τον γνωστό Pat the Cope Gallagher, εδώ, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ισλανδία. Λέγεται The Cope γιατί έπρεπε το όνομα της οικογένειάς του να ξεχωρίσει από άλλες οικογένειες Γκάλαχερ του Ντόνεγκολ και γιατί Κόπ, γιατί ο ε, παππούς, προπάππος του είχε ξεκινήσει ένα συνεταιριστικό πρόγραμμα στην περιοχή. Κάτι το οποίο νομίζω ξεκίνησε με πολύ καλή επιτυχία, ιδιαίτερα στο τομέα της Ελίας και τα λοιπά, αλλά έχει πάρει και άλλες διαστάσεις, ε, όπως και η Credit Union έχει ξεκινήσει συνεταιριστικά. Άρα, λοιπόν, μπορούμε ίσως να κοιτάξουμε λίγο την ιστορία του 21ου αιώνα και τα συνεταιριστικά κινήματα και να διδαχθούμε από αυτή τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Επίσης πιστεύω ότι στην Ευρώπη η ιδέα της αδελφοποίησης, όχι μόνο για πόλεις, αλλά και για σχολεία, νοσοκομεία και το καθεξής, αλλά και συνεταιριστικά ε, σωματεία που ε, έχουν τη δυνατότητα της συνεργασίας. Είχαμε στην Ιρλανδία, παραδείγματι, ένα συνεταιριστικό ε, εργοστάσιο, γεωργικό εργοστάσιο που ε, είχε πάρει πολύ μεγάλο μέγεθος στην Ιρλανδία, το κρατούσαν οι γεωργοί και μάλιστα ξαναγύρισαν στην συντηριστική μορφή πρόσφατα γιατί ήταν ότι αυτό αποδίδει περισσότερο. Το ίδιο βλέπουμε στην Αιθιοπία με ένα συνεταιρισμό που διαθέτει το σπόρο μιας ε, ποικιλία πατάτας κατάλληλης για το κλίμα και τις δαφικέ συνθήκες εκεί και όταν έχει την παραγωγή του ο ο ε, παραγωγός σαν αποζημίωση, σαν τίμημα δίνει στο συνεταιρισμό δύο σακιά σπόρο πάλι που θα πάνε σε κάποιον άλλο παραγωγό και τώρα σιγά σιγά έχει πάρει τις διαστάσεις σε αυτή που χρειάζεται το συνεταιρισμό και για τη διάθεση στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Γκαλέρα. Ε, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τι, τι πιστεύει για αυτό στις δυνατότητες αδελφοποίησης των ε, συνεταιριστικών οργανώσεων της Ευρώπης με αυτές του αναπτυσσόμενου κόσμου γιατί εκεί μπορούμε να προσφέρουμε πολύ μεγάλη βοήθεια, πολύ περισσότερες από ό,τι φανταζόμασταν γιατί μπορούμε να δώσουμε ιδέες για την ανάπτυξη της παραγωγής, το εις τους και έχουμε πολλά παραδείγματα από χώρε που τώρα θεωρούνται ανεπτυγμένε, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Ο κύριο Γκέρεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα προς την ε, συντάκτρια της εκθέσεως που εκφραστώ επί τη ευκαιρία να διατυπώσω ένα ερώτημα. Αν την άκουσα αρκετά, την κατάλαβα αρκετά καλά. Ε, λέτε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει τη γνώμη των εκπροσώπων της κοινωνικής οικονομίας. Δεν είπατε ότι πρέπει να τους προσφέρει αρρωγή η υποστήριξη. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά ισχυρά τα κινήματα αυτά και ότι δεν χρειάζονται ε, υποστήριξη. Ιδιαίτερα από το χώρο της μικροχρηματοδότησης, εκεί όπου αρκεί να λάβει κανείς τεχνογνωσία για να προχωρήσει. Γιατί η μικροχρηματοδότηση νομίζω είναι ένα μέσον που αποδεικνύει πόσο πιο ταπεινός μπορεί να προχωρήσει και να ε, φέρει αποτελέσματα εκεί που κάποιοι πιο μεγάλοι του χρειάζονται πιο σοβαρή υποστήριξη. Παράδειγμα, η αναχρηματοδότηση του συστήματος της μικροχρηματοδότησης περνάει μέσα από τις διεθνείς κεφαλουχικές αγορές και φτάνει σε πολλαπλάσια επιτόκια, μέχρι 15-16% που είναι κατωτετριμένο για τις ε, ε, επιχειρήσεις αυτές που λαμβάνουν την μικροχρηματοδότηση, ενώ το 1,25 στην Ευρώπη ως επιτόκιο δανεισμού θεωρείται ήδη καταχρηστικό ή πολύ ε, βαρύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νικόλα Τέιλορ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η πολυ βαρυ καλωσορίζει την έκθεση. Είναι σημαντική η θεματολογία της. Και εμείς μπορούμε πιστεύω να τη δούμε υπό το φως και της πρόσφατες εκθέσει της Παγκόσμιας Τράπεζας για την απασχόληση των νέων στην Αφρική, Το καθιστά απόλυτα σαφές ότι μοντέλα οικονομικού μετασχηματισμού που γνωρίζαμε στον 20ο αιώνα δεν έχουν πλέον πολύ μεγάλη ε, απήξη στα όσα λαμβάνουν χώρα στην ε, Αφρική και ειδικότερα την υποσαχάρια. Ε, είναι μεγάλη εξάρτηση από το γεωργικό τομέα των νέων για την απασχόλησή τους, αλλά και αντίστοιχα την οικονομική ευμάρεια. Άρα, όπως προγραμμίζει και η Παγκόσμια Τράπεζα, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης περιοχών όπως αυτές για να επιτρέψουν τη βελτίωση των οικονομικών δικών για όλους τους κατοίκους εκεί. Η ορολογία της κοινωνικής οικονομίας όντως δεν είναι πολύ παρούσα στον σχεδιασμό και την ορολογία ή στον διάλογο, ακόμα και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι όλοι είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε χείρα βοηθείας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία αναφέρεται ρητά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ρίζες δημοκρατίας και την ε, αηφόρο ανάπτυξη, όπου λέμε ότι θα πρέπει να αναπτύξει σχέσεις εξωτερικές η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινωνία των πολιτών και ρητά ε, λέει ότι θα πρέπει να ε, υποστηρίξει εταιρικές σχέσεις που υποστηρίζουν κοινωνικές επιλογές, επιλογές κοινωνικής οικονομίας. Επίσης όμως και πέραν αυτού υποστηρίζουμε πολύ αυτό που ονομάζεται άτυπη οικονομία, με την έννοια και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της, κοινωνικής, και της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τον καθένα, με την ε, πτυχή της κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης σε μια παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν οφείλω να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια, πρώτα, μια πρόσκληση για εκδήλωση προσφορών με το πρόγραμμα «Επενδύουμε στον άνθρωπο» Investing in People, που θα επιτρέψει σε παράγοντες της ε, κοινωνικής οικονομίας να συμμετάσχουν και να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Πέραν αυτού, θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει μια προπαρασκευαστική δράση υπό τον κοινωνισμό για την ε, ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και τη θέσπιση ε, επιχειρηματικότητας για την Ανατολική Αφρική. Αυτό είναι προπαρασκευή φέτος και βέβαια θα θέλαμε την υποστήριξή σας στην ε, προώθηση αυτού του τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Γκαλέρα η οποία θα απαντήσει σε τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Δυστυχώς ε, εδώ βρισκόμαστε μόνο σε ένα διερευνητικό πεδίο, είναι διερευνητική έκθεση. Ε, θα, εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε τι πρέπει να γίνει. Σαφής περιορισμός ε, της ε, μελέτης μας είναι ο ορισμός της κοινωνικής οικονομίας, γιατί επικρατεί μια μεγάλη σύγχυση ακόμη και στην, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πολλοί είναι εκείνοι, είτε παράγοντες που δραστηριοποιούνται, είτε ακόμη και αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, που μπερδεύουν την κοινωνική οικονομία με άλλες δραστηριότητες, πράγμα το οποίο βέβαια δεν βοηθάει καθόλου. Το είδαμε άλλωστε και ως πρόβλημα που εντοπίστηκε στη συνεργασία μας και με τους Αφρικανούς ερευνητέ. Δεύτερον, δεδομένα αξιόπιστα για την κοινωνική οικονομία στην Αφρική που θα μας βοηθούσαν να αξιολογήσουμε και να αναγνωρίσουμε τη σημασία του τομέα αυτού δεν υπάρχουν ή ελάχιστα μόνο. Πάντως, πολύ σημαντικό βρίσκω, εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από όλα, βρίσκω το να υποστηρίξουμε την αναγνώριση της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή αναγνώριση των διαφόρων οικογενειών που εντάσσονται σε αυτήν. Είτε πρόκειται για ε, αλληλοβοηθητικές, είτε πρόκειται για συνεταιριστικές οργανώσεις ή άλλους τύπους. Υπάρχουν μελέτες βέβαια στην Ευρώπη οι οποίες αναλύουν το ρόλο, το δυναμικό, τον αντίκτυπο των συνεταιρισμών στον 20ο αιώνα. Και μάλιστα σας καλώ να επισκεφτείτε την ε, ιστοσελίδα του Eurexem, του Ινστιτούτου μας, και να ε, μελετήσετε κατεβάζοντας από το διαδίκτυο αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει σε συνεργασία με, την, ε, με την εταιρική σχέση για, την, ε, για τους συνεταιρισμούς. Είναι πολύ πιο ανθεκτική σε περιόδους ε, κρίσεως η συνεταιρισμοί, πολύ πιο ανθεκτική από μια ε, κερδοσκοπική εταιρεία. Επίσης, ε, η δικτύωση αυτής της εποχής κρίσεως έχει πολύ μεγάλη σημασία να υποστηρίξουμε, να προσφέρουμε εξήγηση για την επιτυχία των πρωτοβουλειών κοινωνικής πρωτοβουλίας, κοινωνικής οικονομίας και έχουμε αποδείξει ότι τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα μοντέλων κοινωνικής οικονομίας ήταν η σε τοπικό επίπεδο εταιρικέ σχέσεις μεταξύ διαφόρων φορέων εμπλεκομένων σε δραστηριότητες αναπτυξιακές. Και εν τέλει, στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο νομίζω είναι να αναγνωρίσει την κοινωνική οικονομία. Μιλώντας για διαβούλευση, Κυρίως είχα στο μυαλό μου αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, αφρικανικά κράτη που θα ήταν καλό πιστεύω να έχουν τακτικότερη επικοινωνία με τους διάφορους τομείς της ε, κοινωνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, δεν έχω πάνω να σας ευχαριστήσω για τη μελέτη σας. Θα αποτελέσει για την προσεχή θητεία πηγή έμπνευσης ασφαλώς. Και τώρα παίρνω στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης για να ακούσουμε την έκθεση μιας αποστολής αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, στην περίοδο 25 με 27 Μαρτίου. Πρόκειται για μια αντιπροσωπεία υπό την συνάδελφα Φιώνα Χόλ, που ήδη η κυρία Χόλ, και ο κύριος Αγκουστίν Διασδεμέιρα, Γκαρσία Κοσουέγα. Έχετε το λόγο κυρία Χολ. Ευχαριστώ πολύ και καταρχάς ζητώ συγγνώμη που δεν έχω καταρτήσει τη γραπτή έκθεση ακόμη αλλά είμαστε ακόμη στη φάση της ε, προετοιμασία. Δεν είχα την ευκαιρία να το συζητήσω με τον κύριο Διασδεμέιρα ακόμη. Έχουμε το θέμα της μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει, το ταχύτερο δυνατό θα σα θα διαθέσουμε το γραπτό κείμενό μα. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι περιμέναμε αρχικά τη συμμετοχή και του κύριου Κάρσμαρεκ αλλά οι αρχές του Σουδάν δεν μπόρεσαν να ετοιμάσουν την θεώρηση του διαβατήριου του εγκαίρους, εγκαίρος, πράγμα το οποίο είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Γιατί στις επισκέψεις, στην επισκέψη αυτή στο Σουδάν και σε πολλές από τις συναντήσεις που είχαμε με εκπροσώπους των Εθνών Εργονοσμών, ακούγαμε διαρκώς παράπονα ως προς την δυσκολία σε σχέση με τις Σουδανικές αρχές ε, για διεκπαιρέωση θεμάτων όπως αυτό της θεώρησης διαβατήριου. Δηλαδή φαίνεται ότι προσπαθούν να ε, παρεμποδίσουν την ε, είσοδο στη χώρα κάποιων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και ήταν πολύ καλό το ότι πήγε το Κοινοβούλιο. Ένα-δύο γεγονότα, στοιχεία τα οποία έχουν ε, πολύ μεγάλη σημασία νομίζω και καταδεικνύουν την γέννη κατάσταση στο Σουδάν. Το γεγονό ότι ο πρόεδρος Μπασίρ έχει παραπευθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραμένει παρόν σε κάθε συζήτηση, δράση αλλά και σκέψη από ό,τι φαίνεται της ε, κυβέρνησης. Ένα άλλο θέμα που έχει φέρει μεγάλη αλλαγή στο Σουδάν. Έχει πειράσει πολύ το Σουδάν την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα που το είχα επισκεφθεί τελευταία φορά το 2004, είναι το γεγονός ότι είναι πια διαφορετικό κράτος το, το νότιο Σουδάν. Έχουν χάσει δηλαδή 75 με 80% από τα έσοδά τους, τους πετρελαϊκούς πόρους. Και ενώ Διαπιστώνουμε βέβαια ότι οφείλεται η ίδια η Σουδανική κυβέρνηση για πολλέ από τι δυσκολίε που αντιμετωπίσει. Το γεγονό ότι έχει χάσει όλους αυτούς τους πετρελαϊκ... όλα αυτά τα έσοδα από του πετρελαϊκού πόρου, από τα οποία εξαρτώταν ε, προφανώ ε, πολύ, έχει πολύ μεγάλη βαρέτητα. Είχαμε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα ε, στι ημέρε τη επίσκεψη. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους τη κυβερνήσεω, υπουργού δηλαδή, εκπροσώπου τη Εθνοσυνέλευση αλλά και εκπροσώπους ε, κυβερνητικών φορέων όπως ε, η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας, αλλά και από την άλλη πλευρά είδαμε εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, διεθνούς βεληνικούς, όπως ε, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και μια άλλη σειρά εκπροσώπων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με πιο μικρές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μια σειρά, ε, είχαμε και μια συνάντηση με νομάδες βοσκούς. Έτσι λοιπόν, είχαμε μια εικόνα από τις επαφές μας με την Σουδανική κυβέρνηση και ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα που λάβαμε από όλους τους υπόλοιπους. Το μήνυμα της Σουδανικής κυβέρνησης και όπως είπα έχουν σοβαρό ε, περιορισμό και στενότητα λόγω της απώλειας των πετρελαϊκών πόρων. Ε, ε, χαρακτηριστικό λοιπόν του ήταν ότι θα μας ζητούσαν περισσότερα χρήματα. Σε οικονομικό επίπεδο ζητούσαν ή επεσήμαναν, επεσήμαναν τριών ειδών προβλήματα, τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ που ανάγονται στην δεκαετία του 90, όπου είχαν προσφέρει καταφύγιο στον Οζάμα Μπιλάντεν οι Σουδανοί, και αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερε είναι οι τράπεζε που δεν δανείζουν στο Σουδάν χρήματα λόγω αυτών των κυρώσεων. Γιατί βέβαια ακόμη και οι τράπεζε από χώρε τη Μέση Ανατολή διστάζουν πλέον, δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ένας, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και πάντα κάπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα τα οποία αντιτάσσονται στην ε, χώρα και Το ζήτημα επίση τη ε, αποχής από τη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της παραπομπής στο ποινικό δικαστήριο του Μπασίρ και ω εκ τούτου το Σουδάν δεν δέχθηκε να υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, άρα έχει αποκλειστεί από εκεί. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει μεγάλη δημιουργικότητα και φαντασία ως προς την ανάπτυξη μέσων υποστήριξης και προγραμμάτων παρόλες αυτές τις, παρόλες αυτούς τους ε, περιορισμούς από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, από, ε, Ευρωπαϊκό Διαρθωτικό Ταμείο, όχι Αναπτυξιακό Ταμείο, συγγνώμη, από άλλα μέσα επίσης που είναι διαθέσιμα. Και τρίτο πρόβλημα, η χώρα έχει πολύ μεγάλο εξωτερικό χρέος. Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο να βρει τράπεζες που θα τις δανείσουν, λόγω της πολύ κακής αξιολόγησης επιστολιπτικής ικανότητας ε, τα, spreading, τα επιτόκια δανεισμού είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχουν προσπαθήσει να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση ε, χρέους με βάση τις αρχές που αφορούν τις ε, υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Αλλά αν αυτό, το, εάν αυτό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε πολιτικό επίπεδο παραμένει αμφίβολο, εδώ σας περιγράφω τα επιχειρήματα της Σουδανικής κυβέρνησης. Αυτά μας είπαν όλοι όσοι συναντήσαμε, όσους συναντήσαμε. Το μήνυμα πάντως από όλους εκείνους που δεν ανήκαν στην κυβέρνηση ήταν πολύ διαφορετικό και πρέπει να πω μας συγκλώνησε. Εμείς είχαμε επισκεφθεί το 2004 τον Ταρφούρ με την Επιτροπή Ανάπτυξη, εγώ προσωπικώ, πριν από 10 χρόνια. Δεν μας είχαν, ε, αυτή τη φορά δεν μα επέτρεψαν να μπούμε στον Ταρφούρ και να το επισκεφθούμε. Ε, Ούτω ή άλλω δεν μα επέτρεψε το Κοινοβούλιο, αλλά και η κυβέρνηση του Σουδάν δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μα δώσει τη σχετική άδεια, διότι η πολιτική τη κυβερνήσεω είναι να περιορίσει όσο το δυνατόν την πρόσβαση στο Νταρφούρ. Οι διεθνεί οργανώσει χρειάζονται άδεια ειδικοί για να κινηθούν εκτός του χαρτούμ, άδεια η οποία μπορεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο ανάλογα με την περίπτωση, με επιχείρημα ότι δεν είναι σωστό το πρόγραμμα ή δεν είναι κατάλληλες οι προθέσεις τους ή αρμόζους ε, η διαδρομή ή ότι υπάρχουν περιορισμοί ασφαλείας για μια συγκεκριμένη περιοχή ή ότι μπορούν να μπουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά θα χρειαστεί να λάβουν την άδεια από τις τοπικές αρχές όταν φτάσουν στην εν λόγω ε, επαρχία και άρα φτάνοντας εκεί βλέπουν ότι τους απαγορεύεται είσοδος. Διάφοροι τρόποι λοιπόν με τους οποίους εμποδίζει την ε, επίσκεψη εκτός του χαρτούμ η κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν δεν μπορέσαμε να πάμε σε κανένα άλλο μέρος εκτός του χαρτούμ, ε, σε κανένα αναπτυξιακό έργο που θέλαμε να επισκεφθούμε, έργα τα οποία είναι κατασκευασμένα και με ευρωπαϊκά κονδύλια. και Ω συνέπεια αυτών των περιορισμών έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο ε, Νταρφούρι στο Νότιο Σουδάν. Πέραν λοιπόν μαζί καλύτερα με αυτή την ε, καταστολή και τον περιορισμό της διακίνησης ε, από τις κυβερνητικές δυνάμεις βλέπουμε και κλιμάκωση της βίας εις βάρος των, τοπικών κοινωνιών. Όταν πήγαμε το 2004 στο Ταρφούρ, η επίσκεψη είχε ακολουθήσει τις, τους μεγάλους εκτοπισμούς, τις, ε, τους εμπρισμούς χωριών και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των χωρικών. Αυτά που μάθαμε τώρα είναι ότι συμβαίνουν ακόμη χειρότερα από αυτά που είχαμε δει το 2003-2004. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ε, ε, έχουν υποχρεωτικά εκτοπιστεί, πολύ περισσότεροι από το 2004. Και η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται τώρα έχει αναπτύξει με μισθοφόρους από την Ιγυρία και το Μαλί, παραδείγματι, μία δύναμη ταχείας ε, ανταπόκρισης η οποία σπέβδει να κάψει χωριά να πυρπολίσει χωριά όπου βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αντίσταση ή αντίδραση για να πιέσει χωρικούς με τον εσωτερικό εκτοπισμό να εγκαταστολιαθούν σε ελεγχόμενους καταβλισμούς. Ο εκπρόσωπος ε, Ρουαντέζος της ε, ε, εκπρόσωπο των ΗΕ σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση μας είπε ότι πρόκειται για εθνοκάθαρση, μας είπε ότι είναι αδύναμη μπροστά στα προβλήματα, ότι οι ίδιοι βρίσκονται υπό επίθεση γιατί μπορούν να κάνουν ε, περιπολίες γύρω από τους καταβλισμούς και να ελέγχουν τα τρόφιμα που μπαίνουν στον καταβλισμό για τους χωρικούς, αλλά έξω από τον καταβλισμό δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τους πολίτες τους χωρικούς. Μας περιγράφει μια κατάσταση δε ε, όξυνσης της, ε, των ε, εκδηλώσεων βίας, των βίων περιστατικών, με συγκρούσεις αντίστοιχες με αυτές του 2004-2003, όπου η κυβέρνηση επιτίθεται όπου βλέπει δυνάμεις ε, αντίδρασης Με πολύ βία η καταστολή Ε, επίσης οι νομαδικοί πληθυσμοί των ε, βοσκών που θα αναφέρω πιο δεξοδικά μετά και γεωργοί άλλοι, γιατί εδώ ήθελα να αναφέρω ότι πρόκειται για παραδοσιακά στοιχεία μένα, αλλά που τώρα έχουν εμπλακεί στον κικαιώνα των εξελίξεων με την κυβέρνηση. Ε, πέραν αυτού, πάντως, βλέπουμε συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων φυλών που και πριν από 10 χρόνια που είχα επισκεφθεί είχαν χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και άρα είχαν πιο ειρηνικέ συνθήκες, αλλά τώρα που η κυβέρνηση δεν έχει τόσο πολλά λεφτά ε, έχουν αρχίσει να αντιπαλεύονται μία την άλλη προσπαθώντας να ελέγξουν φυσικούς πόρους όπως σε μια περιοχή του ε, Νταρφούρ μία φλέβα χρυσού που έχει ανακαλυφθεί. Ε, γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, γενικά υποφέρει σε τεράστιο βαθμό ο πληθυσμός και πάντως η κυβέρνηση δυστυχώς αρνείται τα πάντα, ζει αγνώντας όλη αυτή την κατάσταση και απλώς απαγορεύει να επισκεφτούν τον Ταρφόρ τόσες πολλές διεθνείς οργανώσεις και οργανισμοί. Η, ακόμα και η άδεια του Ερυθρού Σταυρού της ε, Διεθνούς Οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού έχει ανακληθεί γιατί του ζητήθηκε, μάλλον έγινε με την να υποχρεωθεί αυτός να εργαστεί μέσω του, της Σιμισελίνου. Το ίδιο η πατιαρμοστία μπορεί να ασχοληθεί μόνο με ε, πρόσφυγες. Οι εκτοπιστές δεν θεωρούνται πρόσφυγες όμως γιατί είναι εσωτερικός εκτοπισμό ενώ εάν κάποιος προέρχεται από το νότιο Σουδάν ε, δεν, πάλι δεν θεωρείται πρόσφυγας από την κυβέρνηση διότι λογίζεται ως αδελφός Σουδανός και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του, ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Νομίζω ότι αυτά μπορώ να πω προς το παρόν, πέραν μιας σύντομης αναφοράς στους νομάδες βοσκούς. Πάντως, ε, εκτός και αν θέλετε να αναφερθώ πιο διεξοδικά, αλλά ε, με τον κύριο Δίας Δεμέρα πρέπει να πω ότι ανησυχήσαμε πάρα πολύ από αυτά που είδαμε και παρακαλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την πρόταση για το κατεπήγον την επόμενη εβδομάδα για το Σουδάν. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν λαμβάνουν καμία ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή και είναι τεράστια τα νούμερα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος δεδομένου του ότι η Φιώνα τα είπε όλα τα σχετικά με την επίσκεψή μας στις 25-27 Μαρτίου. Να αναφερθώ σε δύο άλλα ζητήματα τα οποία δεν έθιξε η Φιώνα. δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην βοήθεια που τους χορηγείται. Εγώ ίδιος ρώτησα στον Υφυπουργό Οικονομίας για τις ποσότητες που πηγαίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην υγεία και στην ασφάλεια και είπε ότι αγνοεί. Ο αρμόδιος Υπουργός αγνοούσε τα, τα ποσοστά και τις ποσότητες. Ένα κομμάτι λοιπόν της ενίσχυσης ε, πάει για τη χρηματοδότηση των μισθοφόρων, για τη διατήρηση αυτής της εμπόλεμης κατάστασης. Τώρα ένα άλλο ζήτημα είναι το περιβάλλον. Συναντήσαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος ε, και επειδή στη Χαρτούμ ε, υπάρχει, μάλλον από τη Χαρτούμ διέρχεται ο Νίλος, τον ρωτήσαμε για το ζήτημα της ρήπανση των υδάτων του Νείλου. Μας είπε ότι ο Νείλος είναι υγιής, αλλά όταν ρωτήσαμε για την επεξεργασία των ε, λιμάτων ε, ή και των αστικών λιμάτων, μας είπε ότι αυτά τα λίματα ε, δεν ε, τύχαναν επεξεργασίας και οδηγούσαν ε, σε ασθένειες όπως η ελονοσία. Ορισμένα λοιπόν τμήματα του Νείλου ε, είναι μολυσμένα. Το περιβάλλον είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ανησυχητικό, διότι το είδωρα αφενός και η απερίμωση αφετέρου το ζήτημα των ε, ορυχείων στο οποίο αναφέρθηκε η Φιώνα αυτό που είδαμε είναι ότι δεν τηρούνται οι κανόνες προς υπερβάλλοντος κατά την εκτόρυξη. Κάτι ακόμα υπάρχει μια ιστορική διαμάχη ανάμεσα σε γεωργούς και σε κτηνοτρόφους κτηνοτρόφοι, οι ομάδες ε, κτηνοτρόφοι θα πρέπει να μετακινηθούν μέχρι τις αποστάσεις 3.000 χιλιόμετρων με τις οικογένειές τους ε, και γι' αυτό ζητούσαν βοήθεια και ενίσχυση στον τομέα της εκπαίδευσης και της ε, υγείας. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι οι νομάδες είναι δεν είναι ειρηνικά πρόσωπα είναι εξοπλισμένοι, είναι οπλισμένοι και συμμετέχουν στις ε, συγκρούσεις. Τώρα σε ό,τι φορά την κτηνοτροφία θα πρέπει να τα πω στα γρήγορα διότι πρέπει να πάω να ψηφίσω. Η κτηνοτροφία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ε, εγχώριου καθάριστου περιόντος ε, της ε, Αλλά η Ένωση τους ε, βοηθάει, φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει να τους βοηθάει διότι ε, χρειάζεται να διατηρήσει η υγεία των ζώων του ζωικού κεφαλαίου. Πιστεύω λοιπόν πως οι κυρώσεις παρεμποδίζουν τις σχετικές πολιτικές. Νομίζω όμως ότι η έκθεση της Φιώνα είναι πληρέστατη και αντανακλά την πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριο Γκέρντ, το λόγο. Ευχαριστώ. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για την ε, παρουσίαση των δύο εισηγητών ε, που μας μίλησαν για μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση. Τέσσερι παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα η Φιώνα Χόλ μας είπε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη ε, δεν παρεμβαίνει του λόγους ε, που γνωρίζουμε. Αλλά όμως παρεμβαίνει, διότι <clears throat> οι διάφορες διευκολύνσει ε, που χορηγούνται συνέβαλαν σημαντικά στην ασφάλεια των Σουδάν σαν ιδιαίτερα σε ένα κομμάτι του Νταρφούρ. Λοιπόν, υπάρχει εμπλοκή του σχετικού ταμείου, ακόμα και αν ε, είναι λόγω χώρε δεν, δεν θεωρούν ότι λαμβάνουν ε, βοήθεια αναπτυξιακή. Ποιο ενδιαφέρεται για του πληθυσμού, Όλοι λίγο πολύ αδιαφορούν. Η κυβέρνηση η πόλεμοι, η φιλετική δίνουν και παίρνουν και τρίτη παρατήρηση από την ανεξαρτησία η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν. Το νότιο κομμάτι ε, χάρη στις συμφωνίες του 2005 και μετά από το δημοψήφισμα του 2012 ή 2011 καλύτερα Ε, υπάρχει πρόβλημα με τους ε, πετρελαϊκούς πόρους. Ε, το καθεστώς της Χαρτούμ είναι πολύ σκληρό και ανέκαθεν λάβαμε τη βοήθεια της Κίνας στο Ηνωμένα Έθνη. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει και η στάση της Κίνας απέναντι στην Χαρτούμ έχει τροποποιηθεί. Διότι η Κίνα δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον τώρα από το στο παρελθόν. Και παρεμπόδιζε όλες τις κυρώσεις σε επίπεδο ΙΕ. Και υπήρχε πάντα η συνενοχή της Κίνας. Διερωτώμε λοιπόν για αν θα υπάρχει δυνατότητα τώρα να εφαρμοστούν κυρώσεις πιο ευφύης και σε αυτή τη χώρα όλες οι συνδίκες, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην χορήγηση βοήθειας προβλικά είναι αδύνατο να ξεπεραστούν. Μου έρχεται να βάλουν τις κραυγές. Ευχαριστώ πάντως ε, τους ε, δύο συναδέλφους ε, που μας διευκρίνησαν τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να βρούμε κάποιες απαρχές ε, στοιχείων για την επίλυση αυτής της ε, απέσιας κατάστασης. Δεν ξέρω τι όρους θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για την αντικατάσταση που την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει εξωτερική υπηρεσία την οποία εκπροσωπεί η κυρία Δωροθέα Στάρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Δεν την είχαμε πριν από τη συνεδρία, επομένω δεν έχω προετοιμάσει παρέμβαση. Αναφέρω μόνο κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Σουδάν. Συμφωνώ πολύ ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουμε εστιασμένοι στο Σουδάν, γιατί διέρχεται μια κρίσιμη φάση αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή και υπάρχει κίνδυνος αν ε, μπει σε περαιτέρω σύγκρουση, μπορεί αυτό να αποθεροποιήσει ολόκληρη την, ε, την ευρύτερη περιοχή. και για τις περιοχές ε, Ίγκατ και Σαχέλ ε, θα δημιουργηθούν πολύ σημαντικά προβλήματα, για πολλούς λόγους. Ακούσαμε την ε, βία στον για τη βία στον Ταρφούρ ότι έχει φτάσει επίπεδα άνευ προηγουμένου από την γενοκτονία του 2003 και μετά και διεθνείς φορείς δεν μπορούν να, λάβουν πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση στον Ταρφούρ. Υπήρξε μια μικρή ελπίδα με την ανακοίνωση του Προέδρου για την έναρξη δημοσίου διαλόγου. Είναι μια δυνατότητα που πρέπει να αδράξουμε, μια ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε, κατά τη γνώμη μας. Όμως, χρειαζόμαστε πραγματικά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαδικασία που συμπεριλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους και τα ε, οπλισμένα, τις οπλισμένες ομάδες και διάφορες κοινωνικές ομάδες ε, στο Σουδάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση μια τέτοια ε, διαδικασία και εμείς ε, χαιρετίζουμε τις ε, προσπάθειε του αρμόδιου πάνελ υπό την Προεδρία και την ηγεσία του πρώην Προέδρου Τομεμπάκη και του κοινού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ταρφούρ. Και θέλουμε να συνεχιστούν αυτές οι διαδικασίες για την επίτευξη ειρήνης ε, στο Σουδάν. Ε, είπατε κι εσείς ότι είναι δύσκολος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπάρχει και ε, η παραπομπή του Προέδρου στο δικαστήριο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί και καθιστά τον πολιτικό διάλογο πολύ δύσκολο. Όπως θα γνωρίζετε, στην προηγούμενη, την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής δεν συμμετείχε το Σουδάν γιατί θεώρησαν ότι η πρόσκληση που προθύναμε προς ε, τον Αντιπρόεδρο του Σουδάν ε, δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Είναι ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους τέτοιες επισκέψεις είναι πολύ σημαντικές, για να δείξουμε την ευρωπαϊκή παρουσία, να αποστείλουμε μηνύματα, να δείξουμε και στον πληθυσμό του Σουδάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νοιάζεται για αυτούς. Να έχουμε λοιπόν μια παρουσία εκεί και η επίσκεψη αυτή είναι ένα βήμα σε μια σειρά δραστηριοτήτων και ενεργειών του Κοινοβουλίου. Πέρυσι υπήρξε και πρόσκληση του Κοινοβουλίου για νέους, ε, προς νέους ε, πολιτικούς ηγέτες εδώ στις Βρυξέλλες, για μία εβδομάδα νομίζω, για από διάφορα ε, κινήματα και κόμματα και διαμόρφωσαν ε, μια πολύ σημαντική ομάδα που ακόμα και σήμερα έρχεται σε επαφή και μας αποστέλει ε, σημαντικές ε, συμβουλές. υπήρξε και αντιστοιχή πρωτοβουλία προς τα, και προς τα δύο κοινοβούλια. Προς το παρόν όμως έχει τεθεί σε πάυση λόγω των διαδικασιών στο Σουδάν. Αυτά είναι προς το παρόν τα βήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρεντς. Έχετε το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα. Ήθελα να θίξω το ζήτημα των προσκλήσεων που απορρίπτονται από το λόγο λόγω σύστημα, όπως αναφέρετε κι εσείς. Υπάρχει αυτό το ζήτημα που πρέπει να θίξουμε και κλεισμένο το θυρών εφόσον είναι δημόσια αυτή η ανακοίνωση, θα πω ότι θα, γίνουν, θα κάνω παρατηρήσεις και κλεισμένο το θηρόν ε, για το πρόβλημα των ε, προσκλήσεων που αποστέλλονται σε εκπροσώπους ε, χώρες, των οποίων ηγείται κάποιος που έχει παρπευθεί σε διεθνές δικαστήριο. Πρέπει εδώ να επιδείχνουν απαραίτητη δημιουργικότητα και φαντασία, χωρίς ε, να πλήξουμε την αποτρεπτική στάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί αφενός το Σουδάν είναι σχεδόν μια ήπειρος. Δεν εκπροσωπείται στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Είναι κρίμα, γιατί χάνουμε μια σημαντική ευκαιρία να μιλήσουμε με πολύ σημαντικούς φορείς. Ευχαριστώ. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τα καταληκτικά σας σχόλια μέσα σε τρία λεπτά. Η κυρία Χολ, ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, ναι, πράγματι αυτό ισχύει. Ενώ τα κονδύλια αυτά δεν είναι για το πρόγραμμα της χώρας. Υπάρχει ζήτημα για τον DCI και περιφερειακά κονδύλια και ακούσαμε και συγκεκριμένε περιπτώσεις όπου ο εμβολιασμό ε, του ζωικού κεφαλαίου βεβαίω και θα πρέπει να γίνει διασυνοριακά. Και έτσι συμπεριλάβαμε και το Σουδάν στο ε, περιφερειακό πρόγραμμα εμβολιασμού όπως έπρεπε. Μιλήσατε για τον πληθυσμό, συμφωνώ απολύτως. Αυτή είναι η αίσθηση όταν μιλούμε και με την κυβέρνηση ότι δεν νοιάζονται, δεν ενδιαφέρονται για τον πληθυσμό. Υπάρχει μια τρομερή συγκέντρωση εξουσίας σε μια ελίτ στο κέντρο και μετά η περιφέρεια είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι το οποίο απλώς ελέγχουμε. Και δεν υπάρχει καμία πραγματική συμπάθεια ή συμπόνια, αν θέλετε, προς αυτόν τον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε και αυτή τη με της ε, ε, ελάνθρωσης ό,τι αφορά το χρέος. Γιατί ξεκίνησαν αυτή την τεχνική διαδικασία, έχουν μια ενδιάμεση στρατηγική μείωση του χρέους, έχουν και προσωπικό ε, και αντίστοιχες εκθέσεις παρακολούθησης, όμως εμείς δεν είδαμε καμία βούληση να, έχουν, να αυξήσουν τις δαπάνες ε, στην εκπαίδευση ή στην υγεία. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό στον προπολογισμό. Και μας ανησυχεί γιατί υπάρχει και διαφωνία μεταξύ των ε, πρεσβευτών ε, των κρατών μελών. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, είναι, καθιστά πολύ σαφές ότι εκτός και αν υπάρξει κάποια ένδειξη ότι ανοίγονται ε, και θέλουν ε, να ε, βελτιώσουν την κατάσταση για όλο τον πληθυσμό, τότε μπορούμε να το εξετάσουμε. Όμως, είναι ανησυχητική η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το Paris Club και η ΕΠΑ θα πρέπει να συμφωνήσουν. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παρατήρηση για την Κίνα. Αν έχει αλλάξει η προσέγγιση της Κίνας, νομίζω Αν και το περισσότερο από το πετρέλαιο προέρχεται από το, Σουδάν, από το Νότιο Σουδάν, βλέπουμε ότι οι κινεζικέ τράπεζε είναι οι μοναδικές που ακόμα δανείζουν ε, στο Σουδάν. Οι κινεζικέ και μία-δυο στην ε, Μέση Ανατολή. Η Κίνα λοιπόν παραμένει ε, σύμμαχο από ό,τι καταλάβαμε. Και τέλος για τον εθνικό ολοκληρωμένο διάλογο και η ΜΚΟ μας ε, επεσήμαναν ότι δεν πρόκειται καθόλου για τέτοιο ολοκληρωμένο διάλογο που συμπεριλαμβάνει όλους τους φορείς. Ουσιαστικά έχει ως στόχο να ενισχύσει την συνοχή ε, του Εθνικού Κόμματος Υπήρξε λοιπόν μια διαμάχη μέσα στο κόμμα. Προσπάθησαμε λοιπόν, ε, ε, υπήρξε μια προσπάθεια συμφιλίωσης στο ιστορικό του κόμματος. Ποτέ δεν ε, αποτέλεσε μέσο διαβούλευσης μεταξύ πολιτικών ομάδων. Για να έχουμε πραγματικά τέτοιο διάλογο που συμπεριλαμβάνει όλες τις ενδιαφερόμενε ομάδες πρέπει να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό δεν συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόλα για όλες τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει και για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε. Και τώρα το τελευταίο σημείο στην ημερησία διάταξη για απόψε με μια προσωπικότητα πολύ γνωστή που χαίρει τη εκτίμηση τη Επιτροπή μα, όλο κύριο Σόρενσεν, Γενικού Διευθυντή της Γενικής ΕΚΟ, για να συζητήσουμε τα κύρια επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Κύριε Σόρενσεν, ευχαριστούμε θερμά που είσαστε κοντά μας και που δεχθήκατε για άλλη μια φορά να μας επισκεφθείτε για να μας κάνετε για άλλη μια φορά τον απολογισμό των επιτευγμάτων σε αυτή τη θητεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας και να μας δώσετε ίσως και τις προοπτικές και προκλήσεις. Ε, έχετε το λόγο. Έχουμε στη θέση μας περίπου μισή ώρα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ που με δέχεστε, είναι η τελευταία σας από ό,τι βλέπω συνεδρίαση. Άρα μόνο τιμή μπορεί να μου περιποιήσει, αλλά και φιλία να μου δείξει αυτή η χειρονομία. Σε μένα προσωπικά, αλλά και στην ομάδα της ΕΚΟ. Και βέβαια την Επιτροπό μου. Φιλία που μοιράζεται με εσά, αλλά και με όλη την Επιτροπή σας και την ομάδα η οποία εργάζεται άκοπα για να μας προσφέρει την υποστήριξή της. Θα ήθελα να επισημάνω ότι την καθημερινή αυτή στήριξη και αρρωγή την ε, βλέπουμε από πλευρά σας. Κάθε μέρα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τίποτα εάν δεν είχαμε τη δική σας υποστήριξη και αρρωγή. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να σας δώσουμε τις ιδέες μας, τις ε, προτάσεις μας και πρέπει να πω ότι το είδαμε και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν κάποτε διαφορετικές ε, απόψεις ή ότι χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Αλλά, γκρόσο μόντο, αυτή τη θέρμη και την υποστήριξη την αισθανθήκαμε σε όλη μας την πορεία, σε συνεργασία μαζί σας. Και τώρα στα αγγλικά. Ίσως είναι καλύτερο γιατί έχω κρατήσει τις σημειώσεις μου στα αγγλικά, προετοιμαζόμενος για τη συνεδρίασή σας. Και τι ήθελα να πω ότι δεν σκοπεύω να σταθώ στις διαφορές που έχω σχέση με τον προπολογισμό, ιδιαίτερα, αλλά πάντως ήταν και παράξενο να μην αναφερθώ καθόλου στον προπολογισμό. Πάντως θέλω να υπογραμμίσω ότι την υποστήριξη της Επιτροπής σας την ε, αντελήφθη σαφέστατα όταν πήγα στην Επιτροπή των προπολογισμών και υπέστην την ανάκριση του κυρίου Λαμασούρ για διάφορα θέματα. Ε, νομίζω ότι μπόρεσα και να ευαισθητοποιήσω σε μια σειρά από θέματα σε βαθμό που θα μπορούσαμε την επόμενη εβδομάδα να περιμένουμε καλά αποτελέσματα υπό το 150, ένα είδος μεταφοράς δηλαδή από άλλες πολύ σημαντικές γραμμές, ε, από άλλα σημαντικά κονδύλια του προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναπτυξιακή πολιτική και ανθρωπιστική βοήθεια και έτσι θα ήθελα να πω ότι ναι, μεν είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, αλλά ιδιαίτερα θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη προ του συναδέλφου σα για τη στήριξη που μα προσέφεραν και ελπίζουμε να δουν την ανταμοιβή αργότερα με στο χρόνο όταν το προσεχές κοινοβούλιο κληθεί να εξετάσει διορθωτικό προπολογισμό. Μια και υπάρχουν, υπάρχει στενότητα πόρων ως προς τις πληρωμές σε όλο το φάσμα των κονδυλίων. Ε, κάνουμε περικοπές όπου μπορούμε. Αλλά πρέπει να πω ότι πρέπει και οι συνάδελφοι για την, για ανάπτυξη να έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Διότι αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε στη βάση τους τις κρίσεις, τις ε, φυσικές καταστροφές κτλ που είναι και ο σκοπό τη αναπτυξιακή βοήθεια, τότε ναι θα χρειαστεί να εκταμεύουμε διαρκώ χρήματα για να σώσουμε ζωές, αλλά χωρίς προοπτική. Αυτό ελπίζω να το καταλαβαίνουν όλοι στην Επιτροπή σας. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει υπεύθυνη στάση από το προσεχές κοινοβούλιο, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε γιατί θα ήταν μεγάλο σφάλμα να μην προσφέρουμε την υποστήριξή μας σε αυτούς που έχουν ε, υποφέρει τόσο πολύ που και που κινδυνεύουν από τις φυσικές καταστροφές. Επίσης, όχι μόνο εγώ, αλλά και η κυρία Τζορτζίεβα, Κρυσταλίνα Τζορτζίεβα, έχει πιέσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες της, αλλά έχει και η ίδια καταβάλει τεράστια προσπάθεια και έχει δαπανήσει με πολλή ενέργεια. Μπορεί να μην σήμερα εδώ, διότι θέλησε να επισκεφθεί και να υποστηρίξει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τις ισπανικές στη Μαδρίτη, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές περικοπές πόρων και ε, θέλουμε να τους απευθύνουμε το μήνυμα ε, και την παράκληση να συνεχίσουν την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό παρά τους, ε, τις δημοσιονομικές περικοπές να συνεχίσουν όλοι να κάνουν τη δουλειά στο βαθμό που μπορούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Γι' αυτό δεν είναι εδώ η κυρία Τζορτζίβα. Αλλά είναι, αν όχι σώματι, παντός ψυχή παρούσα και μου έχει ζητήσει να διαβιβάσω τους θερμούς χαιρετισμούς της ε, χωρίς λοιπόν αναφερθώ στην, ε, στο κληροδότημα του παρελθόντος θα ήθελα να διευκρίνησω κάποια ζητήματα ότι μπορέσαμε χάρη στη βοήθειά σας και παρά τα προβλήματα να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους το 2012-2013 είμαστε στα 1,35 δισεκατομμύρια ε, νούμερα που είχαμε δει την τελευταία φορά την εποχή του εμφυλίου στη Γιουγκοσλαβία και πάλι δεν είχαμε αγγίξει το επίπεδο αυτό. Δηλαδή ε, βλέπουμε ότι έχουμε ε, αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης έχουμε ξεκινήσει ένα σύστημα, μια μεταρρύθμιση του συστήματος στο επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για τις κατεπίους ανάγκες επίπεδου 3 με το Νότιο Σουδάν, Κεντροαφρικανική ε, Δημοκρατία και Συρία, γιατί έχει βγει από το παιχνίδι το θέμα των Φιλιππίνων, σημαίνει ανάπτυξη μέσω του, συστημά, του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για κινητοποίηση του βέλτιστου δυνατού προσωπικού και άρα υποστήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πρέπει να το έχετε υπόψη αυτό, διότι έχουμε προσωπικό επιτόπου που μπορεί να παρακολουθεί στενότατα τα τεκτενόμενα και έχουμε τη δυνατότητα όταν βλέπουμε τα Ηνωμένα Έθνη να μην τα καταφέρνουν στην περιοχή, να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο και να μιλάμε επευθείας με τη Νέα Υόρκη και τα Ηνωμένα Έθνη και να πούμε κοιτάξτε κάντε κάτι ακόμα είναι αυτό που θα λέγαμε σχέσεις ε, του τύπου όποιος αγαπάει παιδεύει, δηλαδή τους αγαπάμε, τους υποστηρίζουμε, αλλά είμαστε και πολύ απαιτητικοί μαζί τους. Αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα, να έχουμε καλύτερο συντονισμό, ανθρωπιστικό συντονισμό, χωρίς να είναι όλα τέλεια. Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Καλύτερη αξιολόγηση αναγκών, καλύτερη λογοδοσία και ε, λογοδοσία όχι μόνο στο σύστημα αλλά και στον ίδιο τον πολίτη, εκείνον που βρίσκεται σε αυτή την ε, κατάσταση και είναι ευάλωτο. Και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ε, είχα την ευκαιρία να προεδρεύσω της ομάδα χωρικών μπόρεσα προσωπικώ να επισκεφθώ και να συνομιλήσω με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που χωρίς να είναι δημοκρατία είναι πάντω Κονγκό Πρέπει να πω ότι ήταν πολύ ευχάριστο το ότι επισκεφθήκαμε την κόμμα το Μασίση, εκεί που έχουν εκδιωχθεί οι τοπικοί πληθυσμοί και βρισκόνται σε καταβλισμούς. περιοχή όπου 200 τουλάχιστον γυναίκε ενό χωριού έχουν ε, υποστεί βιασμό, τον οποίο οι μισοί τα καν επέζησαν, έχουν σφαγιαστεί και μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μέσω αυτών των προβλημάτων με τι ανθρωπιστικέ οργανώσει, για να δούμε αν πράγματι αυτό που κάνουμε έρχεται στον πολίτη που το χρειάζεται, φτάνει εκεί που πρέπει, αν έχουμε το καταλληλότερο προσωπικό, εάν είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ της, ε, ε, των μονάδων προσφοράς επιστηστικής βοήθειας και εκείνων που προσφέρουν την, ε, τις κουβέρτες Φερρυπίν ή αν είναι ασφαλείς οι γυναίκες όταν χρειάζεται να βγουν από τον καταβλισμό για να αναζητήσουν ε, τροφή, επί παραδείγματι είδωρ κτλ. Γιατί εκεί συνήθως εκδηλώνονται οι βιασμοί. Αν υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση των φίλων όλα αυτά. Και είπαμε, διαπιστώσαμε μετά από αυτή την ε, προσπάθεια, μετά το νότιο, το βόρειο κυβού και, το, και την Κατάγκα, αυτό το τρίγωνο του θανάτου, όπου υπάρχουν ένοπλες ομάδες που καταδυναστεύουν τον τοπικό πληθυσμό και προξενούν τόσα πολλά προβλήματα. Θέλησαμε να δούμε πράγματι αυτό που κάνουμε είναι και το σωστό, εάν φέρνει αποτέλεσμα. Και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή για άλλη μια φορά, γιατί από ε, τα δικά σα χρήματα χρηματοδοτούνται, αλλά είναι οι δικοί μου άνθρωποι επί τόπου και κάνουν καταπληκτική δουλειά, αναπτύσσουν τι προσπαθίε του σε όλο αυτό το πεδίο και την επικράτεια. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που δεν έχει ενδεχομένω εκδηλωθεί 100% αλλά πάντως έχει να κάνει με την διασύνδεση τη ανθρωπιστικής με την αναπτυξιακή βοήθεια. Δηλαδή να ξέρουμε ότι όταν ε, δίνουμε τις οικονομίες μας, όπου τις δίνουμε, η προσπάθεια γίνεται για να ανα προσανατολιστούν τα αναπτυξιακά ταμεία ώστε να ανοίξουν οι βρύσες και να τρέχουν νερό καθαρό, ώστε να ξαναχτιστούν τα σχολεία, ώστε να υπάρχει η βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υποστήριξη για τους ε, πληθυσμούς αυτές τις τόσο ευάλωτες περιοχές. Όλα αυτά έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερη προβολή και πρέπει να πω ότι η διαρκής αυτή πίεση, η διαρκής ε, παρενόχληση των εισαγωγικών από τη δική μας την ε, μονάδα, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη του πολύ καλού συναδέλφους, δείχνει, έχει ε, φέρνει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του ενδιαφέροντος προς τον πιο ευάλωτο και την μετάβαση στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ε, από την ανθρωπιστική βοήθεια στην αναπτυξιακή. Ιδιαίτερα λοιπόν παίρνει μεγάλη σημασία για την υποσαχάρια Αφρική και το Σαχέλ η πρωτοβουλία Αζίγα Σαχέλ Έχουμε επίσης μπορέσει να αναπτύξουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς ώστε να έχουμε ε, συνεργασία και συμπληρωματικότητα, ιδιαίτερα στο κέρας της Αφρικής, τα όσα κάνουμε. Άλλωστε την νότια, τις νότιες περιοχές της ε, Αιθιοπίας, γιατί η Σομαρία είναι πολύ πιο περίπλοκη υπόθεση και διαφορετική, αλλά τουλάχιστον στην Αιθιοπία βλέπουμε ότι έχουμε μοιράσει τα καθήκοντα μεταξύ μας, έχουμε ένα καλό καταμερισμό και προσπαθούμε να εστιαζόμαστε εκεί που έχουμε εμείς πιο ισχυρά πλεονεκτήματα, εκεί που έχουν οι Αμερικανοί, πιο ισχυρή παρουσία ή άλλοι χορηγοί ενδεχομένω και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις επαφές και με τους νομάδες βοσκούς ώστε να εξασφαλίσουν τον βιοπορισμό τους και κάποιες προοπτικές για το μέλλον ή μη τι άλλο. Είναι πολλά υποσχόμενη αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι το, τα, προγράμματα δράσης ε, resilience ε, τα οποία τώρα αναπτύσσονται στην υποσαχάρη Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ έχουν λάβει νέες διαστάσεις. Οι δε χώρες αναπτύσσουν αυτή την αντοχή, το resilience όπως λέμε, στα εθνικά τους ε, προγράμματα. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με επιλογή τομέων και με ε, συνέπεια των έργων. Όταν χτίσετε ένας δρόμος, δηλαδή δεν χτίσετε απλώς ένας δρόμος, εξασφαλίστε ότι η κοινότητες που ζουν γύρω από τον δρόμο αυτό να έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιηθούν για να επισκευάσουν τον δρόμο σε περίπτωση κάποιες καταστροφής, ακόμη και φυσικής με μια πλημμύρα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τους δρόμους, συμβαίνει, και με τα σχολεία. Πρέπει να συνεχίσουν δηλαδή να εργάζονται ακόμη και υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Επαναπροσωνατολισμός δηλαδή της αναπτυξιακής μας δράσης μαζί με την ανθρωπιστική στον τομέα αυτών. Και επίσης Ένα άλλο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ε, οι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη υπόθεση. Οι κυβερνητικέ οργανώσει θεώρησαν ότι θα είχαν ανταγωνιστέ ή ότι θα υποφέρουν τα προγράμματα που τι αφορούν από την παρουσία αυτών των εθελοντών. Εμεί κάναμε μεγάλο κόπο για να τι ότι δεν πρέπει να ανησυχούν και ότι εξασφαλίζουμε μια βάση προσωπικού ε, που θα μπορούσαν από, το οποίο, από την οποία θα μπορούσαν να αντλήσουν ε, υλικό, ε, ανθρώπινο δυναμικό για το μέλλον, νέους που μπορούμε εμείς να καταρτήσουμε και θα έχουν στη συνέχεια, αλλά δεν υπάρχει βέβαια διακρίσεις προς την ηλικία, όπως τελικά αναπτύχθηκε το σχέδιο αυτό τελικά, και από εκεί ο Διεθνής ε, Ερυθρός Σταυρός, το Saving the Children, η UNICEF κτλ. μπορούν να προσλάβουν το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει περάσει από το ασφαλές περιβάλλον στην κατάρτιση. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να του στείλουμε στο καλακάλι σε άλλα μέρη πολύ επικίνδυνα. Αλλά έχουν περάσει μέσα από, έναν, ε, από μια διαδικασία, μπορούν να μάθουν πραγματικά πώ γίνεται αυτή η δουλειά. Ένα άλλο συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι η νομοθεσία για την, για την ε, πολιτική προστασία. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλέ συζητήσει για το πώ ε, μπορεί να ε, συνεργαστεί ο κόσμος της πολιτικής προστασίας με την ανθρωπιστική. Έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε αναζητήσει δυνατότητες για συνεργασία με τους αρμόδιους για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά βέβαια αυτό θα πρέπει να ισχύσει ως με βάση βασικές αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας, ουδετερότητα, βοήθεια προς όλους κτλ. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα σαφέστατο αποτέλεσμα για το πλαίσιο δράσης Γιόγκο που αναμένεται να αναπτυχθεί το 2015 διότι χάρη σε αυτό μπορούμε να έχουμε ένα νομοθέτημα που ήδη έχει τι έχει εφαρμογή σε πολλά κράτη-μέλη. Και μπορούμε να πούμε στον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο, ότι εμεί δεν διεκδικούμε ε, την ε, αυθεντία να υποδείξουμε στου άλλου τι πρέπει να κάνουν, αλλά έχουμε ήδη δοκιμάσει και την ανάπτυξη αυτή τη ε, μονιμότητα και τη αντοχή των έργων και τον τρόπο να περιοριστεί η φτώχεια με τα διαρθρωτικά ταμεία, παραδείγματι. Δεν μπορούμε τώρα να, να επιτρέψουμε τη δαπάνη χρημάτων υπό το, από τα διαρθρωτικά ταμεία, εάν δεν έχει προηγηθεί αξιολόγηση συνεπειών, κινδύνου είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ε, παρουσιάσουμε ως επιχείρημα. Έχει δοκιμαστεί από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης διότι χρειάστηκε να το αξιοποιήσουν. Τώρα μπορούμε να το, να το μεταφέρουμε στον ευρύτερο κόσμο και η Κίνα και άλλα κράτη και μην ξεχνάμε, ε, ε, μην μιλάμε μόνο για τους δρόμους που χτίζονται αλλά ακόμα και για τα εργοστάσια υφαντουργίας του Μπαγκλαντές όπου ξέρετε τα ατυχήματα που έχουν γίνει πρόσφατα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας τρόπος να αλλάξει και η νοοτροπία του κόσμου. Και επίσης έχουμε συνειδήσει και εδώ στρέφουμε λίγο προς το μέλλον του γεγονότος ότι με τις παγκόσμιες εξελίξεις η Ευρώπη θα έχει χαμηλότερο ε, χαμηλό, μικρότερη οικονομική βαρύτητα στον κόσμο και άρα θέλουμε να κινητοποιήσουμε νέους χορηγούς που θα μπορέσουν να ενταχθούν και να υποστηρίξουν το σύστημα. Περίπλοκο όλο αυτό, διότι σε κάθε διαφορετική κουλτούρα και το είπα και άλλη φορά νομίζω στην Επιτροπή σας και νομίζω ότι κάθε κουλτούρα έχει την ε, ιδέα της παροχής βοήθειας των άλλων ε, στον ε, πλησίον, είτε πρόκειται για τον πουδισμό, είτε για το μεθανισμό, είτε για τον χριστιανισμό. Υπάρχει αυτή η έννοια της αλληλοβοήθειας με διαφορετικό μου τρόπο σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε από το σημείο στο οποίο προσφέρει κανείς μια βοήθεια γιατί έχει και πολιτική ιστροβουλία ε, και προχωράει στην παροχή βοήθειας όπως κάνουμε εμείς ανεξαρτήτως της, ε, του χρώματος του δέρματος ε, ή των πολιτικών προτιμήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν, αυτή η μετάβαση είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για πολλές χώρες, αν κοιτάξουμε τις χώρες του Περσικού, όπου οι πόροι βρίθουν, όπου υπάρχουν πολλές οικονομικές δυνατότητες. Αλλά προσφέρονται με πολιτική ιστροβουλία. Και από εμά δεν μπορώ να πω, υπάρχουν κάποιε μη κυβερνητικέ οργανώσει που μπορεί να έχουν πολιτική ιστροβουλία, αλλά πέραν αυτού η οικονομική βοήθεια στηρίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια στηρίζεται στι αρχέ τη ανεξαρτησία και τη ουτερότητα. Πώ το κάνουμε αυτό, πώ έχουμε τι επαφέ με αυτού του ανθρώπου, με το διάλογο. Πάμε στι μεγάλε ανθρωπιστικέ διασκέψει στον Περσικό. Η Κρυσταλίνα είχε πάει στην Διχάτ των Ηνωμένων ε, Αραβικών Εμμυράτων ε, τι προάλλε κάνει τις επαφές. Έχω εξαίρετες σχέσεις με την οργάνωση αραβικών κρατών και τώρα υπό την αιγίδα το, της ομάδας των κυρίων χορηγών. Είμαστε θέση να τους προσκαλέσουμε και να έρθουν να μας μιλήσουν και να συζητήσουμε πώς μπορούν να προσφέρουν καταρχάς, καταρχήν μάλλον την ανθρωπιστική βοήθεια. Βλέπουμε εδώ ότι κάποιοι από αυτούς ανταποκρίνονται Είναι εκπληκτικό το πώ το Κουβέτ, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, αρχίζει να διαθέτει χρήματα στο πολυμερέ σύστημα. Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, πρώτη-πρώτη φορά, χωρί αιρέσει, χωρί προποθέσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά κονδύλα, περνάνε από, από άλλους διάβλους, αλλά πάντως βλέπουμε ότι και εκείνοι ξεκίνησαν σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται ότι είναι προς το συμφέρον όλων. Η Τουρκία, και δεν είναι τυχαίο, το ότι η Τουρκία θέλησε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό ε, συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη για το 2016. Προσπαθώ να κερδίσουν και τη δική τους υποστήριξη για την ομάδα αυτή των ε, χορηγών και πάλι για τον ίδιο λόγο έχουν αυξήσει μαζικά την ανθρωπιστική βοήθεια. Πήραν την ε, Προεδρία λοιπόν. Με την Προεδρία όμως, την Προεδρία ακολουθεί και η η υπευθυνότητα, η κοινή ευθύνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας όρος εκ ε, κάνευ, λοιπόν, για την επιβίωση του ανθρωπιστικού μας συστήματος είναι να κερδίσουμε και να πείσουμε τις χώρες αυτές, και όχι μόνο του Περσικού, αλλά και την ε, Βραζιλία, την, ε, τις Ινδίες, αλλά και την Κίνα βεβαίως, εφόσον θέλουν να παίξουν ένα, ένα πιο ενεργό ρόλο στο παγκοσμίο σκηνικό. Θα περιοριστώ σε αυτά, κυρία Πρόεδρε. Έχω τα διάφορα έντυπα εδώ για την κρίση της Συρίας, ε, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πάει ναι. Είσαστε ενήμεροι, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθώ. Ξέρετε τι είδους προκλήσεις αντιμετωπίζουμε, ενημερωθήκατε. Όπως είπα, μόλις επισκέφθην την ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δεν είναι καθόλου ε, απλά τα πράγματα και καθόλου ευχάριστα. Επισκεφθήκαμε όμως τη χώρα και για να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα βέβαια, αλλά και για να βεβαιωθώ ότι όταν έχουμε να κάνουμε τόσο τεράστιες ανάγκες στη Συρία και τον Νότιο Σουδάν, όπως είδαμε τώρα, και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για να μην αναφερθώ στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τα λοιπά κράτη, ήθελα λοιπόν να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεχάσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικώ εκτοπιστέντων που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται, φαίνεται να είναι η κατάσταση απελπής, αλλά δεν μπορούμε να του εγκαταλείψουμε και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους παρασταθούμε και να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Ακόμη στόχος μου ήταν να αποστείλω ένα σαφέστατο και ισχυρότατο μήνυμα στις, ε, στην κυβέρνηση του Κονκό, τον Καμπιλά και τους υπουργούς του που συναντήσαμε, τον Υπουργό των Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι ο Μουνούσκο θα μείνει, η Μινούσκο, η, επιχείρηση των Εθνών θα μείνει στην ανατολική χώρα, γιατί κοστίζει πάρα πολύ καιρό, ότι δεν θα μείνει λοιπόν επαόριστον. Άρα θα πρέπει να έχει αντιληφθεί ότι άπαξ εξασφαλίσει τη βασική σταθερότητα, θα πρέπει να αναπτύξει τις υπηρεσίες, να λύσει το ζήτημα της ε, ιδιοκτησίας γης και της ε, ε, διαχείριση των ορυκτών, του ορυκτού πλούτου εκεί πέρα, που βρίσκεται σε απόλυτη αναρχία αυτή τη στιγμή, διότι αν δεν το κάνει αυτό ο Καμπυλά και η κυβέρνησή του, τότε θα έχει στα χέρια του τέτοιου είδους φορείς ή αίτια αποσταθεροποίησης και συγκρούσεων που δεν θα μπορεί να τα διαχειριστεί και θα είναι επιπλέον και μόνος του. Αυτά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Για άλλη μια φορά, με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάστηκα μαζί σας και όταν, αρχίσετε, όταν έρθετε, έρθει η ώρα για την ε, προεκλογική σας εκστρατεία, θα έχετε πιστεύω μαζί σας και ένα ε, δώρο από την Κριστίνα Τζορτζίνα που θα είναι, έτοιμο την επόμενη εβδομάδα και μπορείτε και θα είναι βέβαια η αναπτυξιακή αυτή βοήθεια και συνεργασία και μπορείτε να το αξιοποιήσετε με το, με το σύστημα του, της ε, αντιγραφής και επικόλλησης, copy-paste, όλοι σας, με τις φωτογραφίες, με την ουσία, με το υλικό το οποίο εσείς έχετε προσφέρει. Οι αποφάσεις δικές σας είναι αυτές που έχουν φέρει την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια θα υπάρχει και υπογραφή της Κριστέλινα Γεωργίου Ευχαριστώ για την ενημέρωσή σας. Ο χρόνος πιέζεται, πρέπει να βιαστούμε. ο Γκάνος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την υπηρεσία σας, την κυρία Επίτροπο, αλλά και εσάς. Ανέκαθεν μας ενημερώνατε με τρόπο αποτελεσματικό. Έχω δύο θέματα που με απασχολούν και μία ελπίδα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορέσαμε να ε, κάνουμε, να διευθετήσουμε κάπως ε, το θέμα της ε, ανθρωπικής βοήθειας. Νομίζω ότι δεν έχουμε μπορέσει να κάνει κάτι ενώπιον της κρίσης οι οποίες συνεχώς αυξάνονται και παρουσιάζονται. Τι θα πούμε στα τα νέα θύματα στην κεντρική Αφρική όταν, ότι έχουμε μια διαφορά ανάμεσα στις πιστώσεις πληρωμών και στις πιστώσεις υποχρεώσεων. Είναι, είναι παράλογο. Μου είπαν ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφωνήσει σε μια επιπλέον συμπληρωματική χρηματοδότηση. Χρειάζεται να καταβάλουμε παραπάνω προσπάθεια και να κατονομάσουμε τους υπεύθυνους αυτής της κατάστασης. Επειδή βρίσκουμε πάντα κάποιες διαφυγές και κάποια θύματα, θα ήθελα να γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να προχρηματοδοτήσει σε περίπτωση που τα κρατημέλη δεν θα μπορέσουν να προβούν χρηματοδότηση και να καλύψουν την απεχθεί συμπεριφορά τους. Δεύτερον, νομίζω πως ε, σήμερα έχουμε την κατάλληλη ευκαιρία. Είναι η 20η επέτειος από την ε, γενοκτονία στη Ρουάντα. Στην συλλογική μνήμη καταγράφεται ένα ε, έγκλημα κρατικό απόλυτα αψόγως προγραμματισμένο και οργανωμένο. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα από τη γενοκτονία αυτή. Η διεθνής κοινότητα σήμερα είναι καλύτερα εξοπλισμένη και είναι σε κατάλληλη θέση για να προβλέψει και να προκαταλάβει μια νέα γενοκτονία. Αναφέρθηκα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σήμερα έχουμε καταστεί ακόμα πιο ανίκανε για να μην αναφερθώ και στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί στα Ηνωμένα Έθνη τα πιο σημαίνοντα πρόσωπα δεν έκαναν τίποτα. Τότε λιγούρισαν μεγάλες φράσεις και ηλικιότητες, συγγνώμη για τον όρο, και Είδαμε τη δολοφονία 900.000 ανθρώπων σε λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτή τη φορά και κατά λίγο, αυτή τη φορά ελπίζω να μπορέσουμε να οργανωθούμε κατάλληλα για να ασκήσουμε μεγάλη πίεση και έτσι στο μέλλον να μην γελιοποιηθούμε και πάλι όταν θα τεθούν τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κέρενς και ευχαριστούμε που αναφερθήκατε και στο δράμα τη ε, Ρουάντα, το οποίο ακόμα δεν έχει ακόμα κλείσει όπω βλέπουμε. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Μίτσελ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σόρινσεν ε, για την πολύ καλή αυτή παρουσίαση. Εγώ δεν είμαι υπέρ... Δεν, ε, δεν θέτω υποψηφιότητα για επανεκλογή, αλλά Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα ψήφου ε, μετά τι προσπαθίε μου ε, στο μηχανισμό αναπτυξιακή συνεργασία και το καθεξή. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Ότι οι προσπάθειε που έχει γίνει σε τέτοιου είδου επιτροπέ δεν μεταφράζονται, δυστυχώ ε, και από την πλευρά των ψηφοφόρων μας. Αλλάζουν τα πράγματα. Αν αφήσουμε ε, τον ε, αναπτυσσόμενο κόσμο στη μοίρα του, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα και για μας και για τα παιδιά μας. Όμως εδώ βρισκόμαστε για να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα στην έκθεση. πρώτα για τη μείωση των κινδύνων ε, που προκύπτουν από καταστροφές και την ανθεκτικότητα. Εσείς είπατε ότι αυτό μπορεί να σώσει ζωές είναι σαν τη διαφορά μεταξύ peacekeeping και peacemaking, είναι στις ειρήνης ή ε, ειρηνοποιών στοιχείων. Πραγματικά είναι κάτι το ενδιαφέρον αυτό το resilience, αυτή η ανθεκτικότητα και πρέπει να δούμε... Ε, πρέπει να δράσουμε προληπτικά, να μην περιμένουμε δηλαδή να πιάσουμε φωτιά για να έχουμε σταθμό Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στην ΤΕΦΚΟ και πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Και δεύτερον, με όλα αυτά τα τεράστια σκάνδαλα στην Ευρώπη, 23.000 παιδιά χάνουν τη ζωή τους κάθε ημέρα. Και όλα αυτά τα τρομερά στοιχεία που βλέπουμε, ευτυχώς υπάρχει βελτίωση και ευτυχώς έχει σημειωθεί πρόοδος ό,τι αφορά τους ε, στόχους της χιλιετίας, για παράδειγμα. Τώρα βλέπουμε το πεδίο των στόχων ε, αϊφόρων άπτυξης μετά του στόχου χιλιετίας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι σκανδαλώδες το κόστος της έλλειψης Ευρώπης ε, σε ό,τι αφορά την ανταξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Εκπονήσαμε μία έκθεση στις αρχές του χρόνου με τη συνδρομή της ε, Γραμματείας του Κοινοβουλίου για την περισσότερη Ευρώπη και ήμουν εισηγητής. Είπαμε ότι θα σώζαμε, ότι θα εξοικονομούσαμε μάλλον 400 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε δαπάνες ε, συναλλαγών σκεφτείτε τι μπορούσαμε να κάνουμε με όλα αυτά τα χρήματα. Όμως ε, το κύριο εδώ είναι ότι απαιτείται κάποιο είδους διαδρομένη επαφή μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Εθνικών Κοινοβουλίων για να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να αναλάβουν και να πάρουν εξουσίες από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ίσως η Ιρλανδική κυβέρνηση θα πάρει ηγετικό ρόλο σε κάποιε περιπτώσει, η Βρετανική σε κάποιε άλλε. Κάπω έτσι θα πηγαίνει. Όμως πρέπει να το σκεφτούμε, να το επεξεργαστούμε αυτό το ζήτημα. Πώς θα περάσει αυτό το μήνυμα στα εθνικά κοινοβούλια. γιατί μπορούν να συνεργαστούν πιο στενά οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια με τα ευρωπαϊκά όργανα. Αλλά αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, να μας προβληματίσει. Κάτι να κάνουμε σε φορά τη διαρθρωμένη προσέγγιση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή και Εθνικών Κοινοβουλίων για να πιέσουμε το Συμβούλιο να σταματήσει ε, αυτό το φαινόμενο. Ε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στα 6 δις ανά έτος ε, που αναφέρει η Επιτροπή, όμως σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε τα μισά. Αλλά ακόμα και ένα τμήμα μόνο να, κατα... να επιτύχουμε. Φανταστείτε τι διαφορά θα κάνουμε. Πρόκειται για σκάνδαλο και πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Θα ήθελα πραγματικά με ενδιαφέρον να ακούσω τις δικές σας απόψεις και εμπειρίες. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Την ε, κυρία Χο, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ τον κύριο Σόρενσεν για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις. Κατόπιν των όσων ανέφερε και ο κύριος Μίτσελ, θεωρείτε ότι επηρεάζεται και άλλους φορείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για μια παγκόσμια συμφωνία για τη κλιματική αλλαγή, γιατί μιλήσατε για την μείωση ε, των καταστροφών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει διάλογος, ότι έχετε κάποιο είδους επιρροή ε, σε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν μια συμφωνία. Και δεύτερον, με ενδιαφέρουν τα όσα είπατε για τους ε, νέους χορηγούς. Εφόσον πρόκειται κυρίως για μουσουλμανικές χώρες, όπως είπατε κι εσείς, υπήρξαν επικρίσεις ε, για την ανθρωπιστική συνδρομή ότι είναι έτσι πολύ τεχνοκρατικό και ανδροκρατούμενο και έτσι δεν κατανοούμε κάποιες φορές τις ευαισθησίες που υφίστανται. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα χειρότερα στο μέλλον. Θα αλλάξουν οι προτεραιότητες αν οι χορηγοί αυτοί προέρχονται από μια διαφορετική κουλτούρα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Σόρενσεν. Σας λέω από τώρα ότι μετά θα ολοκληρώσουμε την συνεδρίαση και ότι θα σερβιριστεί και ένα ποτό για να αποχαιρετηθούμε. Ο κύριος Σόρενσεν, να πω μόνο ότι δεν ήρθα μόνο για το ποτό, αλλά θα μείνω μετά. Γιατί είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Κύριε Γκέρενς, α, σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσω από τον κύριο Μίτσελ. Κύριε Μίτσελ, πραγματικά κατανοώ τι εννοείτε. Κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και οι πολιτικοί οφείλουν να κάνουν το σωστό. Και αν περισσότεροι πολιτικοί το έπραταν αυτό, τότε ο κόσμος ίσως να ήταν λίγο διαφορετικός. Όλοι λοιπόν έχουμε περιθώριο βελτίωσης, όμως ε, είναι πολύ θετικό το ότι εργαστήκατε για αυτόν τον μηχανισμό αναπτυξιακή συνεργασία, ότι σας απασχολούν τα ζητήματα μείωση του κινδύνου καταστροφών. Ίσως τελικά να μην αντιλήσετε ψήφου από αυτό, αλλά εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Ρωτήσατε εάν καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό τον τομέα, με την ΤΕΦΚΟ, με άλλους φορείς, ε, στο ιστορικό της Επιτροπής, αλλά και με τα κράτη-μέλη. Γιατί ουσιαστικά άπτεται τον όσον είπατε για τα κοινοβούλια, ότι πρέπει να έχουμε επιρροή στα κοινοβούλια, να αναγνωρίζουν ε, ότι και εμεί είμαστε, όπως και εκείνοι, σημαντικοί φορεί, και αν συγχρονίσουμε τις προσπάθειέ μας, είμαστε ανίκητοι, αίτητοι θα είμαστε. Γιατί έχουμε πολλές δυνάμεις του καλού. Τώρα, υπό το θεματολόγιο της ανθεκτικότητας, γιατί εμείς το ξεσηκώσαμε αυτό το ζήτημα, όπως και οι Βρετανοί, κάποιοι Αμερικανοί, αλλά και στη Γερμανία πριν από τις εκλογές. Το καινούργιο στοιχείο ήταν ότι καταφέραμε να αποστείλουμε μια κοινή επιστολή προς όλες μας τις αντιπροσωπείες στις πιο ευάλωτες χώρες, αλλά και σε όλες τις πρεσβείες των κρατών μελών. Επιστολή την οποία υπέγραψα εγώ και ο Φερνάντο από την ΤΕΦΚΟ και όλοι οι γενικοί διευθυντές από όλα τα κράτη-μέλη. Πρωτοφανές αυτό. Και το μήνυμα ήταν, σας παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μας ε, ε, συνάδελφοι, στη Χαρτούμη, οπουδήποτε αλλού, συνεργάζονται από κοινού ε, επί, της, επί τη βάση της ανάλυσης ε, ευαισθησίας, vulnerability analysis, και πώς δρούν για να επηρεάσουν αυτήν την κατάσταση. Τώρα το τι θα γίνει, εγώ Είμαι πραγματιστής, όμως βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η δυναμική. υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συνεργασία και διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις. Δεν θέλω να επιστρέψω σε λεπτομέρειες. Μας απασχολούν ζητήματα από την εκπαίδευση των ε, νέων κοριτσιών ε, στο Νεπάλ μέχρι τους ε, βοσκούς, τους νοτρόφους, πώς πρέπει να σφαγιάζουν κάποια από τα ζώα τους για να επιβιώσει το κοπάδι ε, όταν υπάρχει έλλειψη νερού. Αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε και ένα πρόστιμο πρόσφατα. Εμείς είχαμε πολύ δημιουργικές ιδέες, δηλαδή να αξιοποιήσουμε αυτά τα πρόστιμα για σκοπούς ανθρωπιστικής συνδρομής. Είναι ίσως ανορθόδοξη πρακτική, αλλά ξέρετε, από πολιτικής σκοπιάς εύκολα το κατανοεί κάτι τέτοιο ο πολίτης. Ουσιαστικά συγκεντρώνουμε κάποια κονδύλια, τα οποία μετά διοχετεύονται σε έναν ε, αξιόλογο σκοπό. Οι πολίτες στη Ιδανία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, τα κατανοούν αυτό το πράγμα και κατανοούν ότι δεν μπορεί ένα κρατος μέλος να έχει τον απαραίτητο αντίκτυπο. Γι' αυτό και όλα αυτά που αναφέρατε για τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικά η ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων. Τώρα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, μάλλον όχι. Είναι συλλογική υποχρέωση για όλους μας λοιπόν. Πολιτικοί, πολιτικά κόμματα πρέπει να συμβάλλουν για να υπάρξει σύνδεση μεταξύ του Εθνικού Κοινοβουλίου και των όσων ε, λαμβάνουν χώρα εδώ στις Βρυξέλλες. συμπλήρωσα ένα ερωτηματολόγιο κάποιου Ινστιτούτου για τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης. Και ένα από τα ερωτήματα ήταν πόσο αισιόδοξοι είμαστε. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε πολλά επίπεδα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, για τη σύνδεση των ευρωπαϊκών ε, κομμάτων με τα εθνικά και να υπάρξει ε, λογοδοσία. Επιστρέφω στον κύριο Γκέρενς δεν έχω πρόβλημα να κατονομάσω κάποιον και τις χώρες ε, που ε, μας δυσκολεύουν. Είναι δημόσια όλα αυτά και ούτε μας προκαλούν έκπληξη. Αν πάτε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα τα δείτε όλα αυτά. Τώρα, πιο σοβαρά, λιγότερο με απασχολούν τα 150 εκατομμύρια, γιατί αν ψηφίσει το Κοινοβούλιο, τότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ειδική πλειοψηφία κατά. Η πραγματική δυσκολία θα είναι το φθινόπωρο. Όταν θα έρθει ο τροποποιητικός προπολογισμό που θα αφορά και εμάς και άλλους τομείς πολιτικής. Εκεί θα υπάρξει μια μνημειώδης ε, μάχη, ακριβώς ε, τη στιγμή που θα έχουμε νέα επιτροπή. Το κοινοβούλιο δεν θα είναι τόσο καινούριο, θα είναι μερικούς μήνες ε, μεγαλύτερο λεκιακά. Εγώ ετοιμάζομαι για εκείνη τη στιγμή, γιατί εκεί μπορούν να πάνε πολύ στραβά τα πράγματα. Και αν δεν πάρουμε τα 250 επιπλέον εκατομμύρια που χρειαζόμαστε, τότε θα πρέπει να μεταφέρουμε ένα τεράστιο χρέος που τελικά θα σταματήσει η ανθρωπιστική συνδρομή στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτό είπα και, την και στην Επιτροπή Προπολογισμού την άλλη φορά και τους ε, επειδή τους είπα ότι πραγματικά η Επιτροπή του Προπολογισμού έκανε συστάσεις που όμως απέτυχαν αυτές τις ε, ξακουστές ε, νύχτες του Νοεμβρίου. Δεν ε, πέρασαν λοιπόν και γι' αυτό βρισκόμαστε τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ θα πρέπει να ενημερώσω τον επερχόμενο επίτροπο και να του πω δυστυχώς επτοχεύσαμε. Και δυστυχώ εσεί ω Επίτροπο Ανθρωπιστική Συνδρομή τον πρώτο χρόνο δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γιατί πρέπει να μεταφερθεί αυτό το χρέο. Για τα 250 εκατομμύρια λοιπόν, να είμαι πολύ ξεκάθαρο, είναι απαραίτητα για μα και θα παλέψω μέχρι τέλους για να τα αποκτήσουμε. Για τη Ρουάντα και κατά πόσο έχουμε διδαχθεί κάτι από το παρελθόν. Εδώ πέρα ζυγίζω τα λόγια μου. Όμως ε, στην ε, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία κάποιοι το είχαν προβλέψει πριν συμβεί. Και η Κρυσταλλίνη ήταν ναι, μία από αυτούς. Το έθεσε ε, επικεφαλής της ημέρης της διάταξης, συνεργάστηκε με τους Γάλλους γιατί τα γνωρίζουν καλύτερα, κινητοποιήσαμε πόρους και Υπήρχε όμως το πρόβλημα ότι οι, οι ομάδες μάχης ε, δεν ε, συμμετείχαν. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι και σπάνια θα ακούσετε έναν ε, ανθρωπιστή να ζητά την παρέμβαση του στρατού. Συνήθω θέλουμε το αντίθετο. Όμως, αν δεν μπορεί κάποιος να βγει από την πρωτεύουσα και να, να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια επειδή πέφτουν κεφάλια, τότε χρειάζεται κάποια στρατιωτική ε, παρέμβαση. Τώρα υπάρχει κάποια παρέμβαση, όμως δεν, δεν φτάνει και έρχεται και πολύ αργά. Επομένω, θαύματα δεν υπάρχουν. Με περισσότερες προσπάθειες θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε κάποια στιγμή. Έχει γίνει εσωτερική ανάλυση περιπτώτως για το EIP, αυτά τα δάνεια και τα έχουμε μοιραστεί όλα αυτά με πολύ έξυπνου εκπροσώπους τη επιτροπή, Ακούστε, είναι πολύ καλέ αυτέ τι προτάσει, αλλά δεν πρόκειται να περάσουν. Αυτό είναι το μήνυμα. Όμω εγώ το θίγω συχνά. Γιατί αν δεν μα περνάει με τον έναν τρόπο θα περάσει με τον άλλον. Και έτσι παρουσιάζουμε σε πολιτικό επίπεδο τι ανάγκε μα για την κλιματική αλλαγή και αν βρισκόμαστε σε επαφή με του άλλου. Ναι, υπήρξε αυτή η συζήτηση σε εσωτερικό επίπεδο στην Επιτροπή και ξέρετε ότι υπάρχει ε, σύνδεση μεταξύ μείωση των κινδύνου ε, καταστροφών και ε, μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Ζητούν την εμπρογνωμοσύνη μας όταν πάνε στη Βόνη για να κάνουν αναλυτικό έργο για, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Θέλουν τη βοήθειά μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεργασία όπως ε, υπάρχει και με τους ερευνητές. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλον. Λέτε ότι η ανθρωπιστική συνδρομή είναι κάτι το ανδρικό. Δεν είμαι σίγουρος καθόλου, δεν νομίζω. Πολλές φορές ε, έχουμε ιδιαίτερα γενναίες γυναίκες ε, που ηγούνται αυτών των προσπαθειών και πρόσφατα ήμουν μαζί τους και μπορώ να σας πω να σας τρομερές ιστορίες. Πάνε κάποιοι δηλαδή κάπου με, με τα φορτηγά, μετά σταματάνε εκεί, πάνε με μουλάρια, ξανασταματάνε, πάνε με τα πόδια, εκεί στο τρίγωνο του θανάτου και μετά ε, υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε κάθε χωριό αν μπορούν να αφήσουν εκεί τα φάρμακα και το καθεξής. Μπορώ να σα το πω όλα αυτά, γιατί δεν είναι οι δικοί μου άνθρωποι, είναι άνθρωποι των ΜΚΟ και των διεθνών οργανισμών. Πραγματικά διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Πράγματι, κάποιες φορές όταν ε, μιλώ στην ε, πλευρά της λογιστικής ε, και τεχνικής υποστήριξης, δηλαδή πώς κινούνται τα φορτηγά και τα ολικόπτερα, ναι, πράγματι υπάρχει μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση, όμως χρειάζεται ο συνδυασμό μεταξύ των δύο. Γιατί όλα απαραίτητα είναι. Για τις μουσουλμανικές χώρες, ούτε εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια ανδροκρατούμενη προσέγγιση, όμως βλέπω ότι πρέπει να έχουμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις μαζί τους για να κατανοήσουν την αξία της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας. Γιατί υπάρχει θεματολόγιο, όπως αντίστοιχα ε, και με τις δικές μας ΜΚΟ. Υπάρχει ένα μήνυμα, είτε προέρχεται από τα πάνω είτε από τα κάτω. Πρόκειται ένα έργο εν εξελίξη, όμως πραγματικά πιστεύω στο διάλογο και αν δείτε ε, αυτές τις κουλτούρες στις οποίες ανήκουμε θα, βρούμε, θα βρούμε ομοιότητες. Και αν μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, σίγουρα θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και στηρίζω ε, την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφή. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ακριβώς γιατί ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε δεδομένο ότι αυτές οι αρχές θα υιοθετούνται αυτομάτως από όλους. Όχι, απαιτείται διάλογος για να πούμε ότι εμείς έτσι θα κάνουμε τα πράγματα, εσείς έτσι, πιάνετε πέρα τα κατά και τι θα κάνουμε. Επομένω και η επόμενη Επιτροπή Ανάπτυξη ε, θα έχει πολλά να κάνει. Θα συνεργαστώ μαζί του όπω συνεργάστηκα και με εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Εκεί πέρασε ο χρόνος και δεν έχουμε πια τις μεταφράστριες. Σας που θερμά κύριε Σόρενσεν. And I think it's terribly shocking to know that you are out of money and that we have to make transfer from infrastructure funds or other funds in order to pay for the food and that we are paying for six million Syrians that are